μυστικό πλαίσιο για το διαδίκτυο που καλούμαστε να υπερψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση στο σημείο αυτό. Η θα δεξαχθεί σήμερα. Λυπάμαι για κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και αφήνω τώρα την Προεδρία στον Πρόεδρο κύριο Σούλτς. επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της ε, Επιτροπής σε σχέση με τα συμπεράσματα συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση διεθνών ταμείων και τη συνεδρίαση ηγετών για τις μεταναστευτικές ροές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και την προετοιμασία της διάσκεψης της Βαλέτας στις 11 και 12 Νοεμβρίου του 2015. Ξέρετε κυρίες και κύριοι, την Πέμπτη ως πρόεδρο, την Κυριακή ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου και με πρόσκληση του πρόεδρου της Επιτροπής κ. Γιούνκερ έλαβα μέρος στην ε, διάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για τις μεταναστευτικές ροές των Δυτικών Βαλκανίων. Και όπως είχα δηλώσει από την Πέμπτη, ε, επανέλαβα ότι λόγω της, ε, των τραγικών διαστάσεων της, ε, της κατάστασης ήταν απαραίτητο ο πρόεδρος Γιουνκέρ να συγκαλέσει στις Βρυξέλλες μια σύνοδο όλων των εμπλεκομένων για να ληφθούν αποφάσεις. Ο πρόεδρος Τούσκ και ο υποφαινόμενος απεδέχθημεν την πρόσκληση και λάβαμε μέρος στην διάσκεψη. Πέραν όμως τη διάσκεψη αυτής πρέπει να προσπαθήσουμε να λάβουμε απαντήσεις και αποφάσεις που θα δώσουν μια οριστική λύση στην κρίση, σε διεθνέ επίπεδο. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό το ότι συζητούνται σήμερα εδώ τα πορίσματα των διαφόρων συναντήσεων. Την Κυριακή ήταν απότομα και βία, για να το πω έτσι, ορατό πόσο ανησυχητική έχει μετα... πόσο, πόσο ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει αυτή η κρίση η προσφυγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, στα Δυτικά ε, Βαλκάνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν διάφορους δρόμους για να φτάσουν στην Ευρώπη, που πεινούν, που κρυώνουν, που παγώνουν, που κινδυνεύουν και όπως το είπε και ο Ζων Κλωτιουνκέρ επαπειλείται ανθρωπιστική καταστροφή. Νομίζω ότι το σχέδιο των 17 ε, που αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε στις πρωινές ώρες της Δευτέρας είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί και να τηρηθεί. Ωστόσο, εγώ φεύγοντας από την ε, προχθεσινή συνεδρία, ήμουν πολύ ανήσυχος. Ήταν ε, η ατμόσφαιρα γεμάτη αποφάσματα και φαινόταν να γίνονται, ε, να δίνονται υποσχέσεις που δεν πρόκειται να τηρηθούν. Κυβερνήσεις, δεξιές και αριστερές, που θεωρούν τους εθνικούς εγωισμούς πιο σημαντικούς από τις οριστικές λύσεις, από τις κατάλληλες λύσεις είναι αυτές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την εξέβρεση μιας λύσης στο προσφυγικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό δίνω το λόγο πρώτα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Ντόναλτ Τούσκ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου και τα επόμενα βήματα να πω το ακόλουθο. Η κρίση, οι προκλήσεις ε, που ως Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ενδεχομένω οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. Αναμφίβολα, οι προκλήσεις αυτές θα μπορούσαν να τροποποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε οικοδομήσει. Οι προκλήσεις αυτές θα μπορούσαν ακόμα και να καταστρέψουν κάποια επιτεύγματά μας, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών του Σέγγεν και κινδυνεύουμε ακόμα περισσότερο μέσω των προκλήσεων αυτών να έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό προσκήνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν θα είναι θετικές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι διανύουμε αυτή τη στιγμή εξαιρετικέ περιστάσει, δύσκολε περιστάσει και για αυτέ χρειάζεται ακριβώ να λάβουμε δύσκολε αποφάσει και θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Ω πρόεδρο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θεωρώ ότι και περισσότερο εξημών, θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίσουν την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κοινού πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Δεν θέλω να σκεφτώ αυτή τη στιγμή καμία άλλη εναλλακτική. Εξ αρχής, από το ξεκίνημα της κρίσης αυτής δηλαδή, είχα πει ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλήξει μια συμφωνία για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αλλά τουλάχιστον οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταδείξει ότι η προτεραιότητα είναι η προάσπιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Δυστυχώς όμως η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Όπως είχα πει άλλωστε και στο Κοινοβούλιο εδώ πέρα στην τελευταία μου παρέμβαση, στην προηγούμενη Ολομέλεια. Έχουμε ένα νέο κύμα προσφύγων από το Χαλέπι και από από άλλες περιοχές της ε, Συρίας. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ε, πρόσφυγες οι οποίοι θα φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επόμενες μέρες. Αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι ήμασταν υπέρ μια συμφωνία που θα μπορούσε να συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να χαιρετήσω λοιπόν τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν, ο οποίο επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή τι τεχνικέ λεπτομέρειε αυτή τη συμφωνία. Μια συμφωνία με την Τουρκία θα ήταν ενδεχομένω ε, λογική, θα μπορούσε να βοηθήσει την αναχέτηση των μετασταθετικών αυτών ροών προ την Ευρώπη. Μια τέτοια όμω λύση και συμφωνία δεν θα ήταν εύκολη. Δεν μπορεί καμία τρίτη χώρα, ούτε προφανώ και η Τουρκία, να μα αντικαταστήσει ή να αντικαταστήσει τα δικά μα τα σύνορα. Δεύτερον, Είπαμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν 11 hot spots στην Ελλάδα και την Ιταλία που θα πρέπει να λειτουργούν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η προθεσμία αυτή είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και απαιτεί επιτάχυνση της εργασίας μας, των πόρων μας και του προσωπικού της Frontex, καθώς επίσης και της ΕΑΖΟ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές αυτές υπηρεσίες έχουν το ίμιση του δυναμικού που κανονικά χρειάζονται. Όσον αφορά τώρα τα κέντρα αυτά υποδοχής και ταυτοποίησης, τα hot spots, ξεκίνησε ήδη μια συζήτηση για το πώς θα πρέπει αυτά να λειτουργούν. Είναι ακόμα σε εξέλιξη όμως η συζήτηση αυτή. Τρίτον, συζητήσαμε εκτενώς για το πώς θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τα σύνορά μα, να προασπίσουμε τα σύνορά μα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναλωνόμαστε σε ατέρμονες συζητήσεις ανάμεσα σε αυτούς που είναι υπέρ των ε, ανοιχτών συνόρων και αυτών που θέλουν να υποστηρίξουν τα εξωτερικά σύνορα. Και τα δύο χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε επιτήρηση των εξωτερικών σύνορων για καλύτερη διαχείριση των σύνορων αυτών. Θα πρέπει να σταματήσουμε την παράνομη διέλευση των σύνορων μας. θα πρέπει να καταγράφονται όλοι οι αιτούντε άσυλο και θα πρέπει να οργανώσουμε τα κέντρα υποδοχή. Αυτά όμω από μόνο του δεν πρόκειται να σταματήσουν τη μετασταυτική ροή, αλλά θα τη μειώσουν τουλάχιστον σημαντικά και ω προ αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η Frontex θα αναπτυχθεί περισσότερο πέρα από την φυστάμενη εντολή τη, προκειμένου να μπορεί να παρεμβαίνει και σε συνοριακέ κρίσει με τρόπο πολύ πιο άμεσο και αποτελεσματικό και να λάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά το ζήτημα τη επιστροφή των παράνομων μεταναστών. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όμω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Απότερο στόχο μα είναι η Frontex να έχει τα απαραίτητα μέσα τα οποία χρειάζεται προκειμένου να προσθέσει πλήρω τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει πραγματικά να χαιρετήσω την εξαιρετική εργασία που ε, έχουν κάνει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρηματοδότηση τόσο της Frontex όσο και της ΕΑΖΟ. Παράλληλα όμως θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εσωτερική ελληνική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν να δώσουμε τόσο στην ΑΣ όσο και στη Frontex τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται και να εφαρμόσουμε επίσης τον ε, προσωρινό μηχανισμό μετεγκατάστασης προκειμένου να καταφέρουμε να απαλύνουμε τις χώρες εκείνες οι οποίες επιβαρύνονται περισσότερο αυτή τη στιγμή. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ε, μετανάστευση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με τους πρόσφυγες από την ε, Συρία. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε μία σύνοδο με Αφρικανικούς ηγέτες και Ευρωπαίους προφανώς ηγέτες στην Βαλέτα της Μάλτας. Είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της συνόδου αυτής να καταλήξουμε σε μία εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής όσον αφορά τα ζητήματα της μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν αποφάσισε ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν ισορροπημένα όσον αφορά την αποτελεσματική επιστροφή των παράνομων μεταναστών και τη διάλυση των παράνομων δικτύων διακίνηση μεταναστών. Παράλληλα όμω θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια τη μετανάστευση και θα πρέπει να προωθήσουμε την οικονομική κοινωνική ανάπτυξη τη Αφρική και παράλληλα δεσμευτούμε προκειμένου να δώσουμε και κάποιες νόμιμε οδούς στους νόμους μετανάστες για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ασφαλή κέντρα και υποδομές υποδοχής και θα πρέπει επίσης να δώσουμε βιώσιμε προοπτικέ στους πρόσφυγες και στις οικογένειές τους και μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, μέχρι να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα προελευσής τους, όταν αυτό δηλαδή θα είναι δυνατό. Τέλος, ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να υποστηρίξουν την ύπατη αρμοστία των ΗΕ για τους πρόσφυγες, καθώς επίσης και το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα, καθώς επίσης και να υποστηρίξουν το Περιφερειακό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στη Συρία, καθώς επίσης και το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, θα αναφερθώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έγινε μια προπαρασκευαστική συζήτηση ανάμεσα στου αξιωματούχου του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Υπηρεσία Συμβουλίου ήδη από τον προηγούμενο μήνα. Χαιρετήσουμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κάμερον να θέσει γραπτό τι συγκεκριμένε ανησυχίε του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τι αρχέ Νοεμβρίου. Σα ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Τούσκ. ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιουνκέρ. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κυρίε και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι. Την... Την περασμένη εβδομάδα από τον προσφυγικό δρόμο των Βαλκανίων είδαμε πρόσφυγες ε, να περνάνε από παγωμένα ποτάμια, να κοιμούνται στη λάσπη, στον αέρα. Σε λίγο καιρό πλησιάζει ο χειμώνας, ε, θα τους βλέπουμε στο χιόνι και στην κακουχία. Και ακριβώς αυτή, αυτός είναι ο λόγος κύριε Πρόεδρε που σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο Τούσκ προβλέψαμε την προηγούμενη Κυριακή μία συζήτηση μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών τα οποία δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ε, λόγω της θέσης τους στα Δυτικά Βαλκάνια ε, έχουν ιδιαίτερη σχέση με το προσφυγικό ζήτημα και τους προσφυγικούς δρόμους. Τα οχτώ λοιπόν κράτη με τον Υπουργό των Μεταναστευτικών Θεμάτων από το Λουξεμβούργο και αντίστοιχα των κάτω χωρών ως εκπροσώπους των, ε, της τωρινής και της μελλοντική Προεδρίας. Είχαμε επίσης προσκεκλημένο τον πρόεδρο του Συμβουλίου Τούσκο και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου κύριο Σούλτσο, διότι για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταστεί σαφές ότι αυτή η προσφυγική κρίση δεν αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα κράτη της Δυτικής Βαλκανικής, αλλά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χρειάζεται κατεπίγουσα προσφορά αροχής και δημοσιονομικά για να τηρηθούν οι συμφωνίες και να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που έχει το Συμβούλιο λάβει σε σχέση με τις προσφυγικές, με, το, με την προσφυγική κρίση και χαίρομαι ιδιαίτερα θέλω να το τονίσω που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σε χρόνους ρεκόρ ακολουθήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Υποτροπής και εγκρίνει δίνοντά μας έτσι τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε με έναν ε, συμπληρωματικό προπολογισμό τα μέτρα για την αντιμετώπιση προσφυγικής κρίσης. Ο Αντώνιο Κουτέρες, υπατός εκπρόσωπος για το θέμα της μετανάστευσης, ε, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΑΖΟ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Προστήριξης για το Άσυλο, καθώς ε, και η Σερβία, η Αλβανία, κράτη περιφερειακά ως προς το ζήτημα αυτό, ήταν επίσης προσκεκλημένα. Η πρωτοβουλία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προτίμησε να κάνει αυτή τη συνεδρίαση με τα κράτη δική ε, Βαλκανικής και με ορισμένα συγκεκριμένα κράτη που εμπλέκονται για να δώσει μια πιο λειτουργική διάσταση και να ικανοποιήσει στο ταχύτερο δυνατό διάστημα τις προσδοκίες και προϋποθέσεις των κρατών μελών, αλλά βέβαια και τις ανάγκες των προσφύγων στην υπόθεση αυτή. Εν τέλει, ίσως και να μην χρειαζόταν καν αυτή η συνάντηση. Κανονικά, θα έπρεπε δηλαδή να ήταν μια ομαλή διαδικασία, μια αυτονόητη διαδικασία ότι τα κράτη της Δυτικής Βαλκανικής συνομιλούν και όχι μιλάνε ο καθένας από την πλευρά του και θα έπρεπε όλοι αυτοί που ο καθένας κοιτάει από την πλευρά του να κάνει δηλώσεις να κάτσουν μόνοι τους σε μια ε, τράπεζα διαπραγματεύσεων και να συζητήσουν. Αυτό ζήτησα και εγώ, να συζητηθούν ανοιχτά, ειλικρινά, ειλικρινώς τα ζητήματα, πολυμερός και διμερός. Η επιθυμία αυτή πρέπει να πω ότι σχεδόν κατά υπερβολικό τρόπο ε, υλοποιήθηκε γιατί αυτό που μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας και με τον τρόπο αυτό φάνηκε να παίρνουν διαστάσεις άλλες και να φτάνουν μέχρι υποθέσεις για διάλυση ή για διχασμό με στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ θα έπρεπε κανονικά να συνομιλούμε και να μην είναι εξαίρεση μια τέτοια συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνομιλούν για κοινά προβλήματα. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί αυτό που χρειάστηκε να κάνουμε εμείς την Κυριακή έπρεπε αυτονόητο να είναι για τα κράτη-μέλη και να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς δική μας παρέμβαση. Η συζήτηση ήταν ανοιχτή, ειλικρινής, με εντάσεις σε ένα βαθμό συζήτηση και δεν νομίζω ότι κάθε, από, κάθε μία από τις παρεμβάσεις που ακούσαμε μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παρέμβαση σε διάλογο. Πάντως έγινε η συζήτηση και προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ότι μόνο από κοινού μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς όλους τους παρευρισκομένους γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ότι η Ευρώπη δεν χτίζεται με το να πολεμάει ο ένας τον άλλον, αλλά με το να συνεργάζεται ο ένας με τον άλλον. Η Κυριακή δεν ήταν η μέρα για βαρύγδουπες πολιτικές διακηρύξεις. Ήταν η μέρα για να ανασκουμποθούμε και να συμφωνήσουμε σε ρεαλιστικά επιχειρησιακά μέτρα άμεσης εφαρμογής οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να αντιμετωπίσουν τρεις μείζονες προκλήσεις. Πρόκληση πρώτη. Δεσμεύτηκαν να παράσχουν ε, άσυλο ε, αμέσως ε, σε όλους τους πρόσφυγες, ώστε να μην μένουν στην Ήπεθρο σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Δεσμεύτηκαν να παράσχουν τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ίδρυυση, αποχέτευση, με βοήθεια και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αν αυτό ήταν αναγκαίο. Και χθες ε, η Κροατία ενεργοποίησε το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ζητώντας ε, χειμερινές στέντες, ε, επίσης συσκευές θέρμανσης και κουβέρτες με τον μηχανισμό αυτό τη της Ευρωπαϊκής θα παράσουμε στην Κροατία την απαραίτητη συνδρομή για να βοηθήσει και να περιθάλψει τους πρόσφυγες. Επίσης, θα αυξηθούν οι, κατά 100.000 θέσεις ε, στην Ελλάδα και στα Δυτικά Βαλκάνια οι δυνατότητες υποδοχής και θα ήθελα να ε, ε, επενέσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό που συμφώνησε δημιουργία 30.000 νέων θέσεων απασχόληση μέχρι τα τέλη του τέλους και επίσης ε, ε, την παροχή επιδόματος ενικού για άλλους 20.000. Και επίσης θα ήθελα να επενέσω και τον κύριο Κουτέρες, εκ μέρους της που, που συμφώνησε να ε, αυξηθούν κατά 50.000 οι δυνατότητε παροχή περίθαλψη εκ μέρου τη Αρμοστία στα Δυτικά Βαλκάνια. Συμφώνηθηκε λοιπόν από του ηγέτε ε, να ε, επιβραδυθεί η ανεξέλεγκτη ροή προσφύγων και θα πρέπει η καταγραφή των προσφύγων να γίνουν κατά την είσοδο στα ευρωπαϊκά σύνορα. Επίση θα πρέπει να ενημερώνονται οι πρόσφυγες για τι υπάρχοντες οδού και ποιε θα είναι οι συνέπειε αν αρνηθούν την καταγραφή του. Γιατί αν κάποιος δεν καταγραφεί δεν θα έχει δικαίωμα. Αυτά θα πρέπει να είναι καθαρά και εξάστερα και να τα γνωρίζουν οι πρόσφυγες. Χωρίς καταγραφή δεν νοούνται δικαιώματα, γιατί οι πρόσφυγες έχουν δικαιώματα και ήμουν ανέκαθεν υπέρ των δικαιωμάτων τους, αλλά έχουν και υποχρεώσεις οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στην Ευρώπη. Δεν έχουν μόνο δικαιώματα. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από κοινού σημαίνει και ανταλλαγή πληροφοριών. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε χώρες ε, που έστελναν τους πρόσφυγες από τη μία χώρα στην άλλη ε, και μία χώρα κατηγορούσε την άλλη. Και οι χώρες μιλούσαν η μία για την άλλη, αλλά δεν συνομιλούσαν μεταξύ τους. Αυτή είναι πολιτική πανικού και δίνει την ε, ψευδέστηση της λύσης, ενώ στην ουσία παραβλάπτει τις γειτονικές χώρες και πλήττει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θέλουμε να θέσουμε ένα τέρμα σε τέτοιες πολιτικές. Οι χώρες θα πρέπει να βοηθούν τις γειτονικές τους χώρες με ανταλλαγή πληροφοριών για τις μεταναστευτικές ροές και τις δυνατότητες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στο δρόμο πού έχουν περάσει τα σύνορα, προς τα πού βαδίζουν, πόσες σκηνές, πόσες ε, κουβέρτες υπάρχουν και πώς μπορούν να διατεθούν στις ε, γειτονικέ χώρες που τις χρειάζονται. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό που χρειάστηκε να καταβάλουμε τόσες τεράστιες προσπάθειες για να πείσουμε μερικές από τις δικές μας χώρες μέλη, να ενημερώσουν τις υπόλοιπες χώρες μέλη για τις ε, προσφυγικές ροές που βρίσκονται στα σύνορά τους. Κάτι που για κάποιον ε, φαίνεται αυτονόητο και κοινή λογική χρειάστηκε να συγκαλέσουμε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να πούμε στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να ελοενημερώνονται για τις προσφυγικέ και μεταναστευτικέ ουρέ. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε φόρμα. Θα πρέπει να έχουμε κοινέ απαντήσει σε τέτοια απλά ερωτήματα που ανέφερα. Χθε όλε οι χώρε που ε, ήταν παρούσε στην συνεδρία τη Κυριακή, όρισαν εθνικά σημεία επαφή, αξιωματούχου επαφή για να γίνεται άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει την εφαρμογή αυτή σε εβδομαδιαβάση βάση και ήδη αυτή την εβδομάδα θα έχει μια βίντεο διάλεξη, την Πέμπτη. Οι ηγέτες επίσης συμφώνησαν να ενισχύσουν τη διαχείριση των συνόρων. Και Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη, τα εξωτερικά μας σύνορα και κυρίως μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Φιρόμ και Αλβανίας. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας 400 επιπλέον αστυνομικοί θα αναπτυχθούν στη Σλοβενία. Αυτή τη βδομάδα λέω το, η Frontex θα βοηθήσει στην, την Ελλάδα για την καταγραφή μεταναστών και προσφύγων. Οι χώρες θα εντείνουν τις προσπάθειές τους και μεμονωμένα για να για να επαναπατρίσουν ε, μετανάστες που δεν ε, χρήζουν προστασίας διεθνούς. Και από αυτήν την άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει συμφωνίες επανεσδοχής ε, με χώρες που μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες συμφωνίες και θα συνεχίσουμε το έργο μας για να βελτιώσουμε την εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής όπου υπάρχουν με χώρες όπως το Πακιστάν για παράδειγμα. Ένα άλλο στοιχείο που με εντυπωσίασε ε, ιδιαίτερος παρόλο που το έμαθα πριν ε, ξεκινήσει η συζήτηση αφορά τη συζήτηση για το εξή θέμα. Σχεδόν όλες ε, οι χώρες, χωρίς καμία εξαίρεση, επέσαν την προσοχή μας στο τεράστιο κόστος που έχει η πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την προσφυγική κρίση. Και αντιλαμβάνομαι αυτό το επιχείρημα. Το κατανοώ απόλυτα. Γι' αυτό ακριβώς στις 15 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχω την, την τιμή να προεδρεύω γνωστοποίησε στα κράτη-μέλη ότι όταν θα χαρακτηρίσει τις δημοσιονομικές δαπάνες, τα κονδύλια που θα δοθούν για την προσφυγική κρίση, θα εφαρμόσουμε ευελιξία στην ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας ιδιαίτερα στους, κανόνες, στους αναθεωρημένους κανόνες ε, του Συμφώνου Σταθερότητας, ε, ενισχύοντας το στοιχείο της ευελιξίας στην ερμηνεία τους όποτε προβλέπετε κάτι τέτοιο. Γιατί αντιμετωπίζουμε πραγματικά ένα έκτακτο και σοβαρότατο πρόβλημα. Ένα εξαιρετικό πρόβλημα. Οπότε μπορώ να πω και να διατρανώσω παντού στην Ευρώπη ότι το σύμφωνο είναι σύμφωνο. Το σύμφωνο δεν είναι σύμφωνο όμως με την παλιά του έννοια όταν πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις προσπάθειές μας υπέρ μιας κοινοτικής πολιτικής. Και με βάση την ανάλυση αναχώρα θα δούμε πώς θα ληφθεί υπόψη αυτό, ε, κάτι που δεν έγινε στο παρελθόν, να ληφθεί υπόψη λοιπόν το κόστος ε, της εφαρμογής αυτής της πολιτικής αντιμετώπισης της, της προσφυγικής κρίσης. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν το αναθεωρημένο σύμφωνο και αυτό με εξέταση αναχώρα. Γιατί κάποιες χώρες, ακόμη και από τις μεγάλες, δεν έχουν αρκετές, δεν, έχουν αρκετές προσπάθειες. Αν κάποιες χώρες καταβάλουν εξαιρετικές προσπάθειες, τεράστιες, ε, με τέτοιο πρίσμα θα ερμηνεύσουμε και το σύμφωνο. Αν όμω κάποιε χώρε δεν καταβάλουν τέτοιε σημαντικέ προσπάθειε και δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από το κόστο αυτή τη πολιτική, δεν θα υποφεληθούν από μια πιο ελαστική ερμηνεία του συμφώνου. Αν θέλει κάποιο ελαστική ερμηνεία του συμφώνου, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει ε, επιδείξει την απαραίτητη υπευθυνότητα, το έχει επιδείξει επαρκές αίσθημα ευθύνης. Και αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι περιορισμένος ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόροι μας είναι περιορισμένοι, οι δυνατότητες ευελιξής και ελαστικότητας είναι περιορισμένες και φτάνουμε σχεδόν να αγγίζουμε τα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφίστη προσπαθειών προκειμένου να κινητοποιηθούν όλα τα απαραίτητα δημοσιονομικά κονδύλια και να συγκεντρωθούν ε, στην ίδια προσπάθεια και για τον ίδιο στόχο. Αλλά ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, είναι αρκετά περιορισμένος και δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω τα κράτη-μέλη και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να σκεφτούν τρόπους ε, συμπληρωματικής χρηματοδότησης γιατί κάτι τέτοιο μας χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξαιρετική προσφυγική κρίση. Γιατί είναι εξαιρετική κατάσταση έκτακτη και χρήση έκτακτης χρηματοδότησης. Και στον τομέα αυτό θα ασχοληθούμε, με τον τομέα αυτό θα ασχοληθούμε τις επόμενες εβδομάδες. Η Κυριακή ήταν μια ημέρα ενότητας. Για πρώτη φορά οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων συζήτησαν ε, στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων τα κοινά τους προβλήματα και αποφάσισαν συγκεκριμένες επιχειρησιακές δράσεις για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Τα μέτρα αυτά μάλιστα συμπληρώνουν ε, τα μέτρα που συζητήσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου που σας ε, περιέγραψε προηγουμένως ε, ο πρόεδρος Τούσκ όταν σας ανέφερε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις 15 Οκτωβρίου. Στις 15 Οκτωβρίου λοιπόν και με βάση αυτά που σας είπα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα ένα στόχο. Να επαναφέρω τα κράτη-μέλη για να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν στις 23 Σεπτεμβρίου στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν σημειώθηκε αρκετή πρόοδος και σε μερικές περιπτώσεις ούτε καταδιάνει η πρόοδος που αναμέναμε. Χρειαζόμαστε πρόοδο κυρίως σε δύο τομείς. Πρώτον, θα πρέπει να επιταχύνουμε την εφαρμογή των επιχειρησιακών των μέτρων για να λειτουργήσουν τα κέντρα καταγραφής και οι προσπάθειες μετεγκατάστασης, κάτι που δεν ισχύει μέχρι στιγμής και φυσικά χρειαζόμαστε και δημοσιονομική υποστήριξη διευκρίνησα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις της 23 η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι θεμελιώδους, κεφαλαιόδους σημασίας, αν θέλουμε να εφαρμοστούν ε, οι αποφάσεις που λάβαμε. Τα μέλη του Συμβουλίου είπε ότι θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και τις ε, επικαιροποίησαν κιόλα. Βέβαια, η πρόοδος κινείται με βραδύ ρυθμό, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ταχεία. Τα κράτη-μέλη βραδιπορούν, ενώ θα έπρεπε να αρχίσουν να τρέχουν. Το Σεπτέμβριο τα κράτη-μέλη υποσχέθηκαν να στείλουν εμπειρογνώμονε και να ενισχύσουν τι υπηρεσίε μα. Χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονε στι υπηρεσίε μα, στου οργανισμού μα, κατεπηγόντω για να βοηθήσουμε στην καταγραφή των προσφύγων, να ε, ε, ε, ζητήσουμε δακτυλικά αποτυπώματα και το Ευρωπαϊκό ε, Γραφείο Υποστήριξης ε, ε, του Ασύλου ζήτησε 374 Μέχρι χθε 145 στάλθηκαν. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ακόμη. Επίσης για τους μεθοριοφύλακες της Frontex έχουμε κάποιο πρόοδο. Ζητήθηκαν 775 πυρογνώμονες από τη Frontex. 326 προσφέρθηκαν μέχρι στιγμής από τα κράτη-μέλη. Ωραία, αλλά ιστερεί αυτή η υπόσχεση σε σχέση με την προσπάθεια που απαιτείται. Και για τη μετεγκατάσταση έχουμε κάποια πρόοδο, αλλά όχι αρκετά ταχεία όσο θα έπρεπε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις, να ορίσουν αθηνικά ε, σημεία επαφής και αξιωματούχους επαφής στην Ελλάδα και να κοινοποιούν τις δυνατότητες υποδοχής. 25 χώρες μέλη από τις 26 που το υποσχέθηκαν δεν έχουν ορίσει ακόμη εθνικό σημείο επαφής. Έχουμε για την Ιταλία και μόνο τρεις χώρες ε, όρισαν ε, εθνικά σημεία επαφής για την Ελλάδα. Και εννέα χώρες είπαν ότι ακόμη χρειάζονται 700 υπάλληλοι. Ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε μία απόφαση για επανεγκατάσταση 160.000 προσφύγων. Που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. ενώ, λοιπόν και απόσταση μεταξύ υποσχέσεων και υλοποίησης πρέπει να είναι ως δυνατόν μικρότερο, αλλιώς χάνουμε κάθε είδος αξιοπιστίας. Il ε, Euh, Πριν από τρεις εβδομάδες αποφασίσαμε να διαθέσουμε για τις πολιτικές που τρέχουν και αυτές που θα έρθουν κάθε δημοσιονομικό μέσο που έχει στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο, δημοσιο... ο Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιήθηκε στο μέγιστο. Και στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό η Επιτροπή, αλλά βέβαια είναι χρήματα των πολιτών, των κρατών μελών, θα διαθέσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση της προσφυγικής κρίσης το 2015 και 2016. 4,2 δις γίναν 10 δις επιπλέον για την πολιτική αυτή. Στις 23 Σεπτεμβρίου τα κράτη-μέλη έδωσαν υπόσχεση να συμπληρώσουν τα κενά που παραμένουν. Ωστόσο, στις διμερείς εθνικές συμβολές λείπουν ακόμα 2,3 δις. Για τα κράτη-μέλη μας ε, έχουν μέχρι τώρα δώσει υπόσχεση για 486 εκατομμύρια. Τεράστιο λοιπόν το κενό, το χάσμα. Λίγο πολύ στο δράμα με αυτό που είχαμε από δύο μήνες, πριν από δύο μήνες, 2,3 δηλαδή δις. Πρέπει να γίνουν περισσότερα γιατί κινδυνεύουμε να μην ανέλθουμε σε ύψος των περιστάσεων. Το Νοέμβριο, και το ανέφερα τον όλο μόλις τώρα, ε, ε, προβλέπεται διάσκεψη με τους ηγέτες των Αφρικανικών κρατών, την οποία θέλαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι το πρόβλημα των προσφύγων δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό. Μη σκεφτόμαστε ότι μπορεί να έχουμε από τη μια μεριά τον μεγάλο κόσμο και από την άλλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μέσα στον κόσμο, έτσι το βλέπω εγώ, και πρέπει ως εκ τούτου να δράσουμε σε συνεργασία με τους Αφρικανούς φίλους αλλά δεν θέλω να καταφτάσω εγώ στη Βαλέτα με υποσχέσεις που δεν έχουν τηρηθεί στη Βαλίτσα μου. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο σοβαρό και υπεύθυνο με τους Αφρικανούς ξαδέλφους μας, εάν δεν είμαστε στη θέση να δώσουμε σωστές απαντήσεις σε σχέση με τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Μέχρι τη βαλέτα δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τις τσέπες γεμάτες, όχι με υποσχέσεις, αλλά και με πραγματικές δεσμεύσεις. Και κύριε Πρόεδρε, μια και έχω ξεπεράσει το χρόνο μου κατά πολύ, αλλά το ξέρετε. Δεν θέλω να πω δύο λόγια για την Τουρκία, γιατί προσπαθούμε να ξεκινήσουμε ένα κοινό πρόγραμμα δράσεως με την Τουρκία, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν κατατεθεί, το Συμβούλιο, υπό τον Ντόναλτ Τούσκ τις μελετά όχι μονοτατικά αλλά και με θετική διάθεση. Ο πρώτο αντιπρόεδρος, κύριος Στίμερμανς, έχει αναλάβει τις απευθείας επαφές με την Τουρκία. Χάρη σε αυτόν έχουμε προχωρήσει τόσο. Τον ευχαριστώ θερμά για τις προσπάθειές του, για τις ε, ακαταπόντες προσπάθειε προσπάθειές του. Άλλωστε και τον κύριο Αβραμόπουλο Αρμόδιο για το θέμα των ε, προσφύγων. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω γιατί στρατεύτηκε και εργάστηκε αποφασιστικά στα κράτη αυτά και σε συνεργασία με τα κράτη αυτά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ζητήσω να χειροκροτήσετε για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Επιτροπής ε, δουλεύει, αναλαμβάνει την ευθύνη γιατί διαφορετικά κανείς άλλος δεν το κάνει. Είναι μια καθημερινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα θέλαμε, χωρίς να θέλουν να κανέναν, το ίδιο να κάνανε και οι λοιποί. Να ανασκουμπώνονταν και να δούλευαν εκεί που οφείλουν να δουλέψουν. Και, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει για την υλοποίηση αυτού του κοινού σχεδίου δράσεως να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Το πράττουμε εμείς, το Φραντς Τίμερμανς, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πρέπει όμως και να προχωρήσουμε ταχύτατα. Και πρέπει να πω ότι διαβάζω και σε ένα βαθμό μπορώ να συμμεριστώ τις γραπτές αυτές ε, δηλώσεις και έκφραση επιφυλάξεων, ανησυχιών, ερωτηματικών και προβληματισμών σε σχέση με την υπόθεση αυτής της Τουρκίας. Θα σας πω όμως το εξής. Η Τουρκία στο έδαφος της υποδέχεται 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες πολύ περισσότερα από ό,τι θα τι αναλογούσαν και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ή λέμε της Τουρκίας, στην Τουρκία, κοιτάξτε, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, τα κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεταξύ ημών και ημών Τουρκία έχουμε ανεπίλητα ζητήματα ελευθεριοτυπία, ανθρώπινα δικαιώματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν μας προσφέρει τίποτα στις συνομιλίες με τους Τούρκους συναδέλφους. Ο ίδιος ο Τίμερμανς μπορεί να σας το βεβαιώσει. Γιατί βεβαίω μπορούμε να προσελκύσουμε την προσοχή τη τουρκική κυβέρνηση και των εκπροσώπων τη σε αυτά τα προβλήματα, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με την Τουρκία. Και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε οι πρόσφυγες οι οποίοι τώρα βρίσκονται στην Τουρκία θα παραμείνουν στην Τουρκία και συμφωνούμε ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην ξεκινήσουν προσφυγικές ροές που πάνε προς την Τουρκία να κινούνται προς, τα, προς την Ευρώπη. Εδώ έχει να προσφέρει η Τουρκία κοινωνικές υπηρεσίες στους πρόσφυγες. Πρέπει να φροντίσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι ότι τα παιδιά στην Τουρκία, τα οποία προέρχονται από κάθε χώρα του κόσμου, θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν στο σχολείο. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτοί οι καταβλισμοί για τους πρόσφυγες και να έχουν τα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα του σχολείου για να έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους μετά. Άρα λοιπόν σας αρέσει, σας αρέσει. Είναι βολικό, δεν είναι βολικό. Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες για συνεργασία με την Τουρκία. Τρία δις. Τρία χρειάζεται η Τουρκία για να διαχειριστεί την κρίση. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για κάθε χρόνο προβλέπει 15 με 16 για το 2015 και το 2016 250 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει λοιπόν το υπόλοιπο να το φέρουν τα κράτη-μέλη το υπόλοιπο ποσό, τα 2,5 εκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια που χρειάζονται και που μας λείπουν σε σχέση με το Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου. Πρέπει να συνομιλήσουμε Τουρκία για την ε, απελευθέρωση στο ζήτημα των προξενικών θεωρήσεων, να μιλήσουμε για την ε, νέα κινητοποίηση διαδικασία για την διεύρυνση, χωρίς όμως να οπισθοδρομήσουμε σε σχέση με τις βασικές μας δηλώσει και με τις θέσεις αρχή Και απευθύνω έκκληση προς το σώμα να μας βοηθήσετε, να βοηθήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε δεσμευτικές συμφωνίες με την Τουρκία που θα μας εξυπηρετούν και εμάς ιδιαίτερα, αλλιώς η κατάσταση θα επιδεινωθεί πολύ περισσότερο. Θα προσθέσω επίσης ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να συνομιλήσουμε για το θέμα των κοινών επιθεωρήσεων των ακτών, κοινών ε, δράσεων ακτοφυλακής. Και πρέπει να μιλήσουμε και για προστασία εξωτερικών συνόρων, πρέπει να μιλήσουμε για διαοχέτευση πληροφοριών για τους πρόσφυγες, πρέπει να συνομιλήσουμε για ενημέρωση προς τον πρόσφυγα, όχι τον δικαιούχο ασύλου, προς τον πρόσφυγα ότι θα πρέπει να επανέρχεται στην πατρίδα του όταν έχει διευθετηθεί η κρίση. Ίσως για τη Συρία καθυστερήσει ακόμα αυτό βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε ιδιαίτερα ε, και τα θέματα της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που θα σας ενδιαφέρουν ε, ασφαλώς. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με βάση την επιστολή των πέντε προέδρων στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Θα τηρηθούν οι προθεσμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στα νομοθετήματα. Συνομιλούμε, συζητούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, τα δύο θεσμικά όργανα, όπως άλλωστε οφείλουμε να έχουμε και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε της Επιτροπής, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Πρόεδρος Βέμπερ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όταν ετοίμαζα τη σημερινή μου ομιλία χθες, Είχα αρχίσει να γράφω ναι, είμαστε υπέρ των κέντρων καταγραφής των hot spots, την υποστήριξη, το ασφαλές κράτος προελεύσεως, αλλά τώρα διαπιστώνω ότι την έχω κάνει την ομιλία αυτή αρκετές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο και γι' αυτό ξεκινώ όχι με την αξιολόγηση στα πραγματικά δεδομένα, αλλά με την αξιολόγηση πολιτικής κατάστασης. Διότι διαπιστώνουμε από την συνάντηση Κυριακής ότι θέλει η Ευρώπη να υπάρχει, να αναλάβει ηγετική δράση, να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Αυτό που θέλαμε πάντοτε εμείς. Κατέστη σαφές την Κυριακή. Ο Ζαν Κλωτιούνκερ μας είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε, ότι υπήρχαν πολιτικές δηλώσεις, υπάρχουν προτάσεις νομοθετικές από την Επιτροπή και τον ε, κύριο Αβραμόπουλο, τον ευχαριστούμε θερμά. Ε, σα έχει υποστηρίξει το Κοινοβούλιο σε πολλά ζητήματα, στον προπολογισμό σα έχει στηρίξει και βέβαια η πολιτική μου ομάδα με τα δύο κείμενα, τα νομοθετικά για το ασφαλέ κράτο και για τη μόνιμη υποσώστοση. Σα στηρίζουμε και είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε την ευθύνη να δώσουμε τις πολιτικές απαντήσεις για να μπορέσει η Ευρώπη να, καταστεί, ε, να έχει δυνατότητα δράσης. Για τα κράτη-μέλη τώρα. Θα πρέπει να πούμε κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου ότι δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί. Και θα ήθελα να πω ξεκινώντας πως ελπίζω το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν συζητά και συνομιλεί στο μέλλον να μην φιλοσοφεί γενικά και αόριστα για το μέλλον αλλά να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα και να, γίνονται, να υλοποιούνται οι υποσχέσει που δίνουν τα κράτη-μέλη. Κύριε Τούσκ, εσεί έχετε ω πρόεδρο Συμβουλίου μεγάλη ευθύνη και πρέπει να διαδραματίσετε ρόλο σημαντικό για να δίνονται, ε, να υλοποιούνται οι δεσμεύσει των κρατών μελών. Χρειάζεται να ασκηθεί η πίεση δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να προχωρήσουμε και δεδομένης κυρίως της ε, εποχής που αλλάζει και του επερχόμενου χειμώνα η προστασία του εθνικού κράτους, οι εθνικοί εγωισμοί πρέπει να σταματήσουν εδώ. Η Ευρώπη των Φαράζ και των Λεπέν δεν πρέπει να υπάρχει πια εδώ. Πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις η Ευρώπη. Η Ευρώπη των ε, δεξιών δυστυχώς ε, δεν είναι αρκετά ισχυρή, αλλά δεν μπορεί να δώσει πάνω απ' όλα απαντήσεις και λέμε ότι αν βοηθάει η Ορδανία, αν βοηθάει ο Λίβανος, αν βοηθούν κράτη φτωχά, πρέπει να βοηθήσει και η Ευρώπη. Λέμε ότι η Ευρώπη είναι υπερήφανη και το έχω ξαναπεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι για τα δικαιώματα των χριστιανών μόνο. Και γι' αυτό ο Ντόναλτ Τούσκ πρέπει να Κοιτάξτε, εάν θέλει ισχυρούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, δεν πρέπει να αφήνουμε τον καθέναν να περιμένει στα σύνορα. Με αυτό το πακέτο λοιπόν μπορούμε να υλοποιήσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα. Και θα ήθελα να κάνω και μια κομματική, αν θέλετε, αξιολόγηση κλείνοντας, γιατί αγαπητοί συνάδελφοι ως ΕΛΚ πολλές φορές διαπιστώνω ότι κατηγορούμαστε για τη συμπεριφορά του Βικτόρ Ορμπάν Κοιτάξτε, υπενθυμίζουμε στον ε, Βικτόρ Ορμπάν και το ανθρωπιστικό ζήτημα και εμεί ω ομάδα και το λέω, αλλά πρέπει να επισημάνω εδώ στην Ολομέλεια ότι στο Συμβούλιο των Υπουργών των Εσωτερικών με τον προσδιορισμό των 160.000 ε, κατά την συνεδρίαση αυτή για ποσόστοση προσφύγων, ο Βικτόρ Ορμπάν και τρει σοσιαλδημοκράτε. Ρουμανία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία, Τρία κράτη μεσολυμοκρατικές κυβέρνησεις δηλαδή τάχθηκαν κατά αυτών των ποσοστώσεων. Η Δανία με φιλελεύθερους, ε, οι κάτω χώρε με φιλελεύθερους δεν βλέπουν, να δεν ακούν αυτό που λέει η Άγγελα Μέρκελ ότι πρέπει να κάνουμε την ανθρωπιστική επιλογή και να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα ε, δίνοντας κατάλημα και προστασία στους ανθρώπους αυτούς. Άρα λοιπόν παρακαλώ η κάθε κυβέρνηση να λαμβάνει τις ευθύνες της. Εμείς εδώ ως Ευρωπαίοι πρέπει να φροντίσουμε αυτό το οποίο ε, λέμε να το υλοποιούμε κιόλας. Και αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας ότι έχουμε να κάνουμε με άνοδο των εθνικισμών και των ε, λαϊκισμών αυτών προσπαθούν να εκφοβήσουν τους πολίτες και εμείς έχουμε λάβει μια σοβαρή απόφαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε λάβει μια πολύ σοβαρή απόφαση οι δημοκράτες, οι φιλοευρωπαϊστές συνεργαζόμαστε και δεν επιτρέπουμε στους Ακροδεξιού να επηρεάζουν την νομοθεσία. Αυτό προσπαθούμε, αυτό προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και παρακαλώ και τους λοιπού συναδέλφου από τις άλλες πολιτικές ομάδες να πράξουν το ίδιο και σε επίπεδο εθνικών ε, πολιτικών και κυβερνήσεων για την Πορτογαλία και με κάθε σεβασμό προς τον πρόεδρο της ε, χώρας ε, θα σημειώσω ότι προσπαθεί να μην δοθεί κυβερνητικός φόκος στους ακραίους της αριστεράς της Πορτογαλίας. Αυτό κάνουμε όλοι οι δημοκράτες σε όλη την Ευρώπη και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουμε την πορεία της Ευρώπης στη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα Υπάρχει μια, προφορική, μια ε, μπλε κάρτα, θέλετε να τη δεχτείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο αυτό το οποίο είπατε. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Κογκρέσο του ΕΛΚΑ συνταχθήκατε με μια λαϊκιστική προσέγγιση αυτή του κυρίου Ορμπάν ένας από το κόμμα του μάλιστα εξελέγει και ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Επομένως μην κατηγορείτε τους σοσιαλιστές, μην μας κάνετε μας υπεύθυνου, γιατί οτιδήποτε και να λέτε αυτή τη στιγμή Νομίζω ότι θα πρέπει η έρευνα να γίνει περισσότερο στα πλαίσια των δικών σας των κομμάτων, της δικής σας πολιτικής ομάδας. Μη συνεχίστε σε αυτή τη γραμμή, κύριε Βέμπερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως ε, δεν με καταλάβατε καλά στα ουγγρικά. Να σας το επαναλάβω. Η απόφαση για 160.000 ε, πρόσφυγες που θα πρέπει να καταναμηθούν με δίκαιο τρόπο στην Ευρώπη είχε αντίθετη την ουγγρική κυβέρνηση του Ορμπάν και τρεις σοσιαλδημοκρατικέ. Το επαναλαμβάνω. Είπε ο Ορμπάν ότι δεν είναι καλή αυτή η απόφαση για την Ουγγαρία. Αλλά σας λέω ότι και ο Βίτσο της Σλοβακίας, σοσιαλδημοκράτη και δικός σας εταίρος, είπε ότι θα την εφαρμόσει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σημειώσω αγαπητή συνάδελφοι ότι πρέπει να σταματήσουμε να ρίχνουμε ένα στο φταίξιμο το, στον άλλον, οι δημοκράτε εδώ στο Κοινοβούλιο, για να μην διευκολύνουμε αυτού εκεί τους ακραίους που σα δείχνουμε το δάχτυλο και να μην κάνουμε το παιχνίδι αυτών. Το ίδιο με αυτό που συμβαίνει και στην Πορτογαλία προσπαθούν να αποκλείσουν του ακραίου αριστερού από την κυβέρνηση. Εκ μέρους της ομάδας Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Πιτέλα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σούλτσε, κύριε Γιούνκερ, κύριε Τούσκα. Πραγματικά δεν μπορώ να κρύψω την ανησυχία μου. Το ότι αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες προσπάθειες διχόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι προστρέχουν αυτή τη στιγμή και λένε ότι τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πραγματικά μας ανησυχεί μας ανησυχεί ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά της παγκοσμιοποίησης, κατά του Ισλάμ, κατά του Ισραήλ, κατά της Ρωσίας, κατά των μεταναστών, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μητριάς όπως την αποκαλούν. Όλοι αυτοί οι οποίοι στρέφονται κατά θα μπορούσαμε να τους αποκαλέσουμε ότι ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εξορισμού είναι κατά χωρίς να έχουν αναλύσει καθόλου την κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει πέρα από αυτές τις προσπάθειες διχόνοιας που βλέπουμε να γίνει και μία ανάλυση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά θα κερδίσει τη μάχη όταν όπως είπε και ο κύριος Γιούνκερ και όπως έκανε άλλωστε την Κυριακή, όταν καταφέρει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει συγκεκριμένε προτάσεις όσον αφορά την ε, κατάσταση που πλήγει τις βαλκανικές χώρες. Θα έχει κερδίσει τη μάχη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα είναι σε θέση να δείξει ότι είναι έτοιμη και αυτό το έδειξε άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της, έτοιμη να αναλάβει γρήγορα και αποφασιστική δράση σε έκτακτες καταστάσεις. Θα έχει κερδίσει όμως τη μάχη η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως όταν θα καταφέρει να δείξει ότι είναι πολύ πιο δυνατή από τον ιό αυτό του φόβου και του εθνικισμού και όταν θα καταφέρει δηλαδή να δώσει πιστικές απαντήσεις, να ανταποκριθεί πιστικά και αποτελεσματικά. Κάνω μια έκκληση λοιπόν προς όλες τις φιλο... φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις οι οποίες βρίσκω εδώ, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεξάρτητα από το πολιτικό φάσμα το οποίο πρεσβεύουν να αναλάβουν δράση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσουμε στο κέντρο της δράσης μας τον φίλο ευρωπαϊ... Ε, ευρωπαϊσμό. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήσουν συντρίμια και από την άλλη υπάρχουν άλλοι που θέλουν να προωθήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμα και την ευρωπαϊκή δράση. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να ελοποιούμε όλες αυτές τις αποφάσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Δηλαδή να έχουμε έναν μηχανισμό μετεγκατάστασης των προσφύγων, ο οποίος θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα σύστημα hot spots, κέντρων καταγραφής και ταυτοποίησης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προασπίσουμε το σύμφωνο Σέγγεν, να προασπίσουμε το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών για ελεύθερη κυκλοφορία. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να ανορθώσουμε νέα τύχη, νέα εθνικά σύνορα. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί λύση σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τρίτε χώρε, όπω για παράδειγμα με τι Βαλκανικέ χώρε, όπω αποφασίστηκε στη Σύνοδο τη Κυριακή. Και είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να μην σεβόμαστε τα δικαιώματα των προσφυγών. Όπως είπε ο κύριος Γιούγκερ, αντιμετωπίζονται απλώς ως μια ανθρώπινη μάζα που μετακινείται και σπρώχνεται από τη μία χώρα στην άλλη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τις χώρες οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην προσφυγική κρίση. Το είπε και ο κύριο Γιούγκερ, θα πρέπει να προσαρμόσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και να δείξουμε ευελιξία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μια τέτοια απόφαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να μην υπολογίσουμε στου εθνικού προπολογισμού και στο Σύμφωνο Σταθερότητα τα χρήματα που δίνουν τα κράτη-μέλη για την προσφυγική κρίση. Όσον αφορά την Τουρκία, δεν μπορούμε να αφήσουμε την Άγκυρα μόνη τη να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση στη, Ρησία, θα, στη Συρία. Θα πρέπει πολύ γρήγορα να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο δράση για την Τουρκία. Θα πρέπει όμω να σαφέ ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δώσουμε εμεί λευκή επιταγή στην τουρκική κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης με την Τουρκία αλλά και να προωθήσουμε την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελευθεροτυπίας και των μειονοτήτων στην Τουρκία. Και τέλος, όπως είπε και ο πρόεδρος Τούσκα, προχωράμε σιγά σιγά προς τη σύνοδο της Βαλέτας. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική. Να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε οικονομικά την Αφρική προκειμένου να μειωθούν οι προσφυγικές ροές από την Αφρική. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτόν τον τρόπο. Αυτό το λέγαμε στο παρελθόν. Χρειάζεται μια πραγματική πλέον ουσιαστική εταιρική σχέση με την Αφρική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τι Αφροκανικές δημοκρατίε. Θα πρέπει να ενισχύσει του θεσμού τη Αφρική θα πρέπει να καταπολεμήσει τη διαφθορά, να ενισχύσει το εκπαιδευτικό σύστημα και να υπάρχει μια ισότιμη ροή επενδύσεων και από τις δύο πλευρές. Πολλά πράγματα λοιπόν πρέπει να κάνουμε όλοι μας τα κράτη-μέλη και οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις μας για να επιλύσουμε την κρίση αυτή προτού να είναι πολύ αργά. Και άλλη μια φορά θα ήθελα να αφαιρθώ σε έναν γνωστό Ιταλό ποιητή, και σας ζητώ συγνώμη για την εθνικιστική μου αυτή τάση, όπως έλεγε ο Δάντης. Εδώ πέρα πραγματικά μιλάμε για την αξιοπρέπειά μας. Κύριε Πιτέλα, ο κύριος Χριστοφόρου θέλει να σας κάνει ερώτηση. Συμφωνείτε? Παρακαλώ κύριε Χριστοφόρου. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι συμφωνούμε ότι τα δυόμισι εκατομμύρια προσφύγων πρέπει να παραμείνουν στην τουρκία και σε αυτό το ζήτημα πρέπει να επικεντρωθούμε. όμω ήθελα να ρωτήσω τον κύριο πιτέλα εάν συμφωνεί ότι το προσφυγικό θέμα είναι ένα ξεκάθαρο προσφυγικό θέμα και οφείλει και η τουρκία και όλε οι χώρε να επιδείξουν ευαισθησία και σε καμία περίπτωση αυτό το ζήτημα όπω φαίνεται εκ μέρου τη τουρκία δεν καταντά στοιχείων εκμετάλλευση και εκβιασμού προ την ευρωπαϊκή ένωση για να εξυπηρετήσει άλλου στόχου συμφωνείτε λοιπόν ότι το προσφυγικό για την τουρκία είναι προσφυγικό αλλά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ένταξη εφαρμογή αρχών και αξιών άνοιγμα κεφαλαίου σεβασμού του πρωτοκόλλου της άγκυρας η τουρκία πρέπει να τα εφαρμόσει και να τα υλοποιήσει χωρίς να υποχρεωθεί η ευρωπαϊκή ένωση να υποστεί εκβιασμούς και απειλές εκ μέρους της τουρκίας που όφιλε να στηρίξει την ευρωπαϊκή ένωση στα θέματα του προσφυγικού άλλωστε είναι θέμα ευαισθησίας είναι θέμα ανθρωπιστικής κρίσης που η ε, τουρκία σε καμία περίπτωση με ανήθικο τρόπο δεν έπρεπε να βάζει αυτά τα ζητήματα στην πλάστη. Θα πρέπει να σας πω ότι πλεονάζετε με την παρέμβασή σας, γιατί εγώ είπα σαφώς, σαφέστατα, ότι δεν δεχόμαστε να δώσουμε λευκή επιταγή στην τουρκική κυβέρνηση. Θέλουμε να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, αλλά επί τόπου θα προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ε, ε, ελευθερία έκφρασης και την, το σεβασμό των μειονοτήτων. Άρα δεν απαρνούμαστε τις αρχές μας και τις αξίες μας. Θα πρέπει να εκτελέσουμε το πρωτόκολλο της Άγκυρας και να βοηθήσουμε την Τουρκία στις μεταναστευτικές ώρες, ε, ροές συγγνώμη, Συρίων. Ο κύριος Καμάλ ε, από την Ισιά. Ευχαριστώ πολύ η κρίση των μεταναστευτικών ροών ίσως θα περάσει, θα βγει σε λίγο από, τις, από τα πρωτοσέλιδα αλλά δεν πρόκειται να λυθεί γρήγορα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τα τετριμένα επιχειρήματα αν είμαστε φιλόι αντί Ευρωπαίοι. Υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα και οι άλλοι που πιστεύουν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα. Ας είμαστε σαφείς τουλάχιστον για αυτά που πρέπει αμέσως να γίνουν τώρα να σταματήσουμε να δίνουμε την εντύπωση ότι οποιοδήποτε είναι πρόσδεκτος και να φροντίσουμε να περιθάλπουμε τους πιο όσους χρειάζονται περισσότερο, όσοι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, να σταματήσουμε με μονομένες χώρες να ανοίγουν τα σύνορά τους για να υποχρεώνουν τις υπόλοιπες να τα κλείνουν και να δούμε τι μπορεί να κάνει η κάθε χώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο θέμα μεταναστευτικών ροών και προσφύγων. Υπάρχει κίνδυνος γεωπολιτικής κρίσης στη Συρία. Η σύραξη συνεχίζεται. Η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να αποσταθεροποιήσει τα σύνορα της Ένωσης για να αποφύγει την προσοχή στην Ουκρανία. Με αυτά, σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουμε το, 10, το σχέδιο της Κομισιόν με 10 σημεία αλλά όλα αυτά τα σχέδια που έχουν ακουστεί δεν υποκαθιστούν την δράση. Πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Να δεχτούμε μόνο τους πρόσφυγες, τους πραγματικούς και που έχουν τις περισσότερες ανάγκες και να επιστρέψουν όσοι απλώς θέλουν να εκμεταλλευτούν το κοινωνικό μας σύστημα. Παρόλα αυτά, πρέπει να δεχτούμε όλοι ορισμένους πρόσφυγες. Έχουμε υποχρέωση Μερικές χώρες κάνουν περισσότερα από άλλες βέβαια και μερικές προσπαθούν να κάνουν. Άλλες δορίζουν χρήματα και άλλες απλώς αποφεύγουν το πρόβλημα. Πρέπει όλες οι χώρες να συμμετάσχουν με συντονισμένη δράση και όταν λέω όλες οι χώρες δεν εννοώ μόνο της Ένωσης, εννοώ όλες τις χώρες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συμβολή της Τουρκίας, της Ιορδανίας και του Λιβάνου, αλλά επίσης πρέπει να αναρωτηθούμε πότε θα αναλάβουν δράση οι πλουσιότερες αραβικές χώρες και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι χώρες στα σύνορα της Ένωσης και στα Βαλκάνια πρέπει να ενισχυθούν. Οι έλεγχοι στα σύνορα να ενισχυθούν, αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σταθεροί, αυστηροί. Πρέπει να δηλώσουμε στους μετανάστες, όχι στους πρόσφυγες, ότι πρέπει να περάσουν από τα νόμιμα κανάλια. Έτσι μόνο θα σώσουμε ζωές, αντί να ενισχύουμε τον κόσμο να διακινδυνεύει τη ζωή του. Έχουμε ζήσει γενιές που έζησαν δύο παγκόσμιους πολέμους και αν θέλουμε να διατηρηθεί η ειρήνη και η ευημερία πρέπει κάτι να κάνουμε τώρα, να μην το πάρουμε για δεδομένο. Ο κόσμος αλλάζει. Οι συσχετισμοί δυνάμεων αλλάζουν μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής αλλά μειώνεται η παραγωγή. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και η ιστορία μας δείχνει ότι για να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές προκλήσεις πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί μα σύμμαχοι και ποιοι όχι. Οι γονείς μας αντιμετώπισαν τις προκλήσεις της εποχής τους και τα παιδιά μας θα αντιμετωπίσουν νέες διαφορετικές προκλήσεις. Πρέπει κάτι να κάνουμε λοιπόν και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ή να κάνουμε κάτι ή να καταφύγουμε πάλι στο παρελθόν. Πρέπει να έχουν όλοι ένα μέλλον στην Ένωση. Από τα προγράμματα δράσης να δούμε ποιους πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε. Να αρχίσουμε τη εφαρμογή των ποσοστώσεων και να βοηθήσουμε πραγματικά και τους πολίτες μας και τους ε, πρόσφυγες. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Χρονικά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Απλώς σας ευχηθώ την προσοχή σε αυτό. Γύρω στη μισή ώρα είναι η καθυστέρηση. Όποιος παίρνει το λόγο, σηκώνονται μετά ένα σωρό μπλε κάρτες. Θα ήθελα παρακαλώ να σας πω τι είναι αυτό το σύστημα εξυπηρετεί τη σαφήνεια των συζητήσεων και τη δυνατότητα να κάνει κάποιος μια ερώτηση σε έναν ομιλητή. Διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι σηκώνεται η γαλάζια κάρτα πριν ανοίξει το στόμα του ομιλητής. Δεν έχει νόημα αυτό να αποκτά κανείς περισσότερο χρόνο με το σύστημα της γαλάζιας κάρτα. Κύριε Κόμπορν, θέλατε να κάνετε ερώτηση στον κύριο Καμάλ. Κύριε Κόμπουρν, θέλετε να κάνετε ερώτηση στον κύριο Καμάλ. Ούτε αυτό είναι έκπληξη. Να δούμε, να ακούσουμε με έκπληξη την ερώτησή σας. Κύριε Καμάλ, δέχεστε την πλακάρτα. Ευχαριστώ, πρόεδρέ μου. Κύριε Καμάλ, ο μόλος ε, τρόπος να ελέγξετε τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι συγκεκριμένος. Πώς ε, εσείς και ο κύριος Κάμερον θα καταλάβετε ότι ο μόνος τρόπος ελέγχου των σύνορων είναι φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε άλλο τρόπο να το κάνετε εκτός αυτού. Καμάλ, χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούσατε τον κύριο Σούλτς για το νόημα της μπλε κάρτας θα μπορέσετε να πείτε ό,τι θέλετε κατά το δημοψήφισμα και μην ξεχνάτε ότι μια συγκυβερνητική κυβέρνηση που πρόθεσε το δημοψήφισμα, όχι εσείς που φωνάζετε από τις άκρες. Εκτός μικροφώνου. Για τους φιλελευθέρους τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω Καλό είναι να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες ενδοβρετανικές συζητήσεις και ανταλλαγές για το βρετανικό δημοψήφισμα. Ναι, εντάξει, χειροκροτήστε, χειροκροτήστε. Μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο που θα ήθελα να πω στο Μάρφετ Βέβερ είναι ότι δεν πρόκειται εδώ για καλυστία ή διαγωνισμό, Μάρφετ, η προσφυγική κρίση μεταξύ ε, φιλελευθέρων, σοσιαλιστών ή χριστιανοδημοκρατών. Δεν είναι καλυστία ούτε διαγωνισμός. Έτσι κι αλλιώς πάντα χαμένοι θα είμαστε. Γιατί αν έχετε στο πλευρό σας τον Όρμπαν που είναι ο σκληρός και τη Μέρκελ που δείχνει συμπόνια, πάντα θα κερδίζετε και πάντα δίκιο θα έχετε. Η πραγματικότητα λοιπόν δεν είναι διαγωνισμός μεταξύ μας, αλλά μεταξύ των εθνικιστών και των λαϊκιστών που θέλουν να καταχραστούν αυτή την κρίση για να καταστρέψουν την Ευρώπη και να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι ο ανταγωνισμός, όχι μεταξύ μας λοιπόν. Ας σταματήσουμε να αλληλοκατηγορούμεθα και να αυτή η κυβέρνηση η ΟΤΑΔΕ και ο ΔΗΝΑ. Το πρόβλημα είναι οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Αυτό έδειξε ο Ζαν Κλοντ Κιούνκερ σε 25 λεπτά μέσα. Και τον ευχαριστώ που το έπραξε με έναν τρόπο πάρα πολύ λεπτομερή. Τι έκανε. Παρέθεσε ένα μακρύ κατάλογο αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Εδώ και μήνες τώρα είτε πρόκειται για τη μετεγκατάσταση. Δεν έχουν γίνει αρκετά. Τι γίνεται με τον προπολογισμό, πάλι δεν έχουν γίνει αρκετά. Και όταν πρόκειται να αποσταλούν ε, δημόσιοι υπάλληλοι για τον ε, έλεγχο των συνόρων και πάλι δεν γίνεται. Το πρόβλημα δεν είναι εδώ μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο μπορεί να λυθεί και να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα. Αυτό έχουμε σήμερα απέναντί μας. Και εδώ είμαστε ενωμένοι. Δεν υπάρχει λόγος να ε, πολεμάμε ένα στον άλλον, γιατί ποιος υποφελείται, αυτοί εκεί πίσω με τις μπλε κάρτες ε, που θέλουν να επιτίθενται στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, γιατί είναι υπαρξιακή αυτή η κρίση. Μια κρίση υπαρξιακή που μπορεί να ξεπεραστεί μόνο ε, εφόσον βασιζόμαστε στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Τούσκ, τώρα αποφάσισε το Συμβούλιο να το καταλάβει ότι χρειάζεται έλεγχο στα σύνορα με ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα φρούριο, αλλά μαζί Ελλάδα, Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία να ελέγχουμε τα σύνορα, να καταγράφουμε τους πρόσφυγες, να φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις για τη διευκόλυνση των ανθρώπων και να ζουν εκεί σε καλές συνθήκες και όχι τις εικόνες που έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Εκεί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά εμείς ανάμεσα σε εκείνους ε, που είναι οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες να γίνει διάκριση. Και εκεί θα οργανωθεί η μετεγκατάσταση. Παρακαλώ κύριε Τούσκ, έκκληση σα απευθύνω. Ξέρω ότι δεν φταίτε εσεί το Συμβούλιο φταίει, αλλά τουλάχιστον στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στη Σύνοδο να αποφασίσουν για αυτή την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή, διότι δεν υπάρχουν τα ελληνικά σύνορα ούτε τα βουλγαρικά είναι ευρωπαϊκά, είναι ε, ε, ταυτόχρονα γερμανικά, βελγικά, ολλανδικά, γολικά. Ε, είναι κοινά σύνορα όλα αυτά, δεν είναι μιας χώρας. Εκεί θα πρέπει να το αποφασίσετε. Για να σταματήσει αυτός ο δρόμος των Βαλκανίων, όχι στα Βαλκάνια, είναι στα σύνορα της Βουλγαρίας, της Ελλάδας. Εκεί θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτά τα ευρωπαϊκά ε, σώματα ακτοφυλακής και σύνοριοφυλακής που να είναι διεθνή να ασχολούνται με την καταγραφή και την επανεγκατάσταση. Και ό,τι σας προτείνω. Μην τους κάνετε χριστουγεννιάτικο δώρο στο Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Εάν δεν μπορούν να αποφασίσουν τώρα, για το κοινό σύστημα ασύλου που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και ε, το κοινό σύστημα οικονομικής μετανάστευσης που επίσης χρειαζόμαστε γιατί πολλοί γνωρίζουν ότι πολλοί καταχρώνουν αυτού του συστήματος τελικά ασύλου για να έρθουν ως οικονομικοί μετανάστες στην Ευρώπη. Αυτό είναι το διακύβευμα. Το Δεκέμβρη που είναι σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Μην τους κάνετε χριστουγεννιάτικο δώρο, μην πάνε διακοπές, να τους πιέσετε, να τους κρατήσετε εκεί μέσα ε, στο κτίριο αυτό το κτίριο που είναι η έδρα του Συμβουλίου αυτό τον καιρό και είναι το ευρωπαϊκού τύπου οικοδόμημα. Ξέρω κύριε Τούστ ότι είστε υπέρ εσείς. Θα πάρτε μια απόφαση επιτέλους. Πάρτε μια απόφαση να δώσετε εντολή στην κυρία Μογκερίνη να αρχίσει πρωτοβουλίε στο δικό της επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην πηγή της κρίσης. Κανείς δεν το αναφέρει αυτό. Ποια είναι η πηγή. Είναι η συνεχιζόμενη σύραξη στη Συρία Χρόνια ολόκληρα καθόμαστε και γυρνάμε από την άλλη με σταυρωμένα τα χέρια και θέλω ότι βλούμε. Θα πρέπει να δώσει το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εντολή στη Μογκερίνη να εμπλακούμε ως Ευρώπη, εξ της Ευρώπης. Γιατί το θεωρώ εξωφρενικό και έσχος. Στη Βιέννη, ήσασταν παρούσα πριν από λίγες μέρες κυρία Μογκερίνη, στη Βιέννη, ε, στη Βιέννη, στην καρδιά, στο κέντρο της Ευρώπης, συνεδριάζουν για τη Συρία. Και ποιο είναι εκεί. Η Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Αμερική και Ρωσία, η Ευρώπη απούσα τουλάχιστον στο συνέδριο της Βιέννης το 1815 ήμασταν γύρω από το τραπέζι. Αυτή τη στιγμή που είναι και 21ος αιώνας απουσιάζουμε ενώ συμβαίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ερήμην μας όλα αυτά. Όπως και με τις Αζόρες. Θυμάστε που είχε διοργανώσει ο κύριος Μπαρόσο για το Ιράκ. Επίσης απούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Καλά δεν ήταν καρδιά τότε, ήταν περιφέρεια. Ας δώσουμε λοιπόν εντολή στην κυρία Μογκερίνη και παρακαλώ αξιοποιήστε τη πλήρω. Να ανοίξετε τις πόρτες ε, έστω και βία σε αυτές τις συνεδριάσεις για να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε φαγόφστατ. Περιέργως ο κύριος Έθριτς έχει ερώτηση, υποθέτω, για εσάς. εσάς. Yeah. Κύριε question. Ναι, θέλω μια αποσαφήνιση από τον κύριο Φερχόφσταντ. Είπατε ότι εμείς που ζητάμε συχνά μπλε κάρτες είμαστε κακοί άνθρωποι γιατί εμποδίζουμε τις συζητήσεις και είμαστε εναντίον όλων. Κι όμως εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη μετανάστευση. Εμείς δεν είμαστε κατά των πάντων. Απλώς είναι μερικοί από εμά που είναι υπέρ της συζήτησης και της δημοκρατίας και της ελευθερίας, είμαστε όμως κατά της Ένωσης και όσων εκπροσωπούν εσείς και οι φίλοι σας. Γι' αυτό υπάρχουν οι γαλάζιες κάρτες και είναι τόσο σημαντικές. Εγώ δεν έχω τίποτα κατά των γαλάζιων καρτών, αφού είναι μπλε όπως το χρώμα της ομάδας μου. Δεύτερον, δεν έχω τίποτα εναντίον τους γενικότερα. Εσείς όμως συνεχώς κουνάτε γαλάζιες κάρτες και λέτε ότι αντιδράτε στα πάντα. Συνεχίστε, συνεχίστε. Μ' αρέσουν οι γαλάζιες κάρτες σας. Δεν είπα τίποτα. Από την Ιωτική Αριστερά το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ιγκλέσιας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την πρώτη φορά που παρενέβην εδώ ήταν 15 μήνες πριν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να σας παρουσιάσω το πολιτικό μου κόμμα και να μιλήσω στο Κοινοβούλιο. Τότε είπα ότι θέλαμε μια διαφορετική Ευρώπη, μια Ευρώπη που να μην είναι τόσο σκληρή με τους αδύναμους και όχι τόσο συγκαταβατική με τους ε, έχοντες εξουσία. 15 μήνες μετά ισχύει η ίδια κατάσταση. Τότε, πριν 15 μήνες, μίλησα για τους Ισπανούς μαχητές που καταπολέμησαν το φασισμό, κάτι το οποίο ήταν η καλύτερη συνεισφορά της χώρες μου για την Ευρώπη, για μια Ευρώπη κοινωνική, δημοκρατική που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν ακούω τους ξενόφοβους σήμερα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εκείνοι ε, που τους εκφόβησαν είπαν τον «Ο Πασαράν» και δεν δέχομαι να ακούω αυτή την υποκρισία από αυτούς που χύνουν κροκοδίλια δάκρυα και που μιλάνε για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Βέμπερ, μιλήσατε για άκρα. Ε, λάβετε υπόψη τι συνέβη στην Πορτογαλία. Να ξέρετε ότι πολλές φορές οι πολίτες ψηφίζουν διαφορετικά από αυτό που εκφράζετε εσείς ο εκπρόσωπος των φιλελευθέρων θα μου ζητήσει συγγνώμη γιατί 15 ε, μήνες αφού κοιτάει τον εαυτό του στον καθρέφτη δεν, ε, ε, προσπάθ, δεν κατάφερα εγώ να προφέρω το επίθετό του. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι τα βασικά στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής τα πληρώνουμε σήμερα με την ταπείνωση και τη μιζέρια που ζουν χιλιάδες οικογένειες στις πύλες της Ευρώπης. Μιλάμε για πολέμους και για κατάπτωση της Ευρώπης σε ε, ανθρώπους που αντιμετωπίζουμε με σειρματοπλέγματα. Μην ξεχνάμε τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει ε, αυτή η κατάσταση, η εμπόλεμη κατάσταση και η φτώχεια. Δεν μπορούμε να ταπεινώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτό σημαίνει ότι ταπεινώνουμε την Ευρώπη. Γιατί το ίδιο σημαίνει, κύριε Βέμπερ, όταν τελειώνουμε με την ευημερία, με τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, να δίνουμε τις ε, κυβερνήσεις τα μεγάλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα και να παραδίδουμε τη δική μας εξησία. Και εσείς κύριε Γιούνκερ ως ε, Υπουργός Οικονομικών κάνατε συμφωνίες με μεγάλες ε, πολυεθνικές έτσι ώστε να έχουν σχεδόν μηδενική φορολογία ενώ οι φορολογούμενοι της Ευρώπης ε, πλήρωναν τους φόρους τους. Και εσείς κύριε Ιούνκερ καθόσαστε εδώ και εσείς κύριε Πιτέλα γιατί εσείς οι σοσιαλιστές είχατε μία μεγάλη συμμαχία με, τους, με το ΕΛΚ. Και κύριε Πιτέλα θα πρέπει να σταματήσετε με αυτή την επονίδη στη μεγάλη συμμαχία και μεγάλο συνασπισμό επιστρέφω στη χώρα μου για να μην πια υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς στις κυβερνήσεις. Αλλά πριν φύγω θέλω να σας πω κάτι. Σταματήστε με την πολιτική σας. Η κρίση των προσφύγων δεν λύνεται με σύρματοπλέγματα, με αστυνομία. Δεν μπορείτε να παίζετε σκάκι με τους λαούς της Μεσογείου βοηθήστε την ειρήνη και αυτούς που φεύγουν από μια κατάσταση τρόμου. Μη συνεχίζετε να καταστρέφετε την αξιοπρέ... αξιοπρέπεια της Ευρώπης, κύριε Γιούνκερ. Από τους Πρασίνους, το λόγο τώρα έχει η κυρία Χάρμς. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε συνάδελφε Βέμπερ, αν θέλετε κάτι να κάνετε πραγματικά σε αυτή την οξία κατάσταση και να συνεισφέρετε για την επικοδομητική λύση, πάρτε τηλέφωνο τον κύριο Ζέχοβερ και να το πείτε. Αντί ε, να κάνει αυτές τις δημόσιες τυμπανοκρουσίες, να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Φράιμαν και την κυρία Μέρκελ για να το λύσουν. Μπορεί να το κάνει αυτό και θα μας χρησιμεύει σε όλους. Καταρχάς θα ήθελα να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Δεν νομίζω ότι ουσιαστικά συζητούμε σήμερα ή θα πρέπει να συζητούμε για βαθιά κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κρίση και ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο σήμερα σοβεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλοί άλλοι λαοί υποφέρουν πολύ περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Και αν δεν σταματήσουμε πρώτα απ' όλα να συζητάμε για τον εαυτό μας, για τις δυσκολίες μας, να ομφαλοσκοπούμε, δεν θα είμαστε σε θέση να συνεισφέρουμε για την επίλυση της κατάστασης στη Συρία και περιοχή ή νοτίος της Σαχάρας ή γενικότερα νοτίως της Μεσογείου για να αλλάξουν κάπως τα πράγματα. Στο μεταξύ πραγματικά τρομακτικό αυτό που βλέπω ε, πόσο εσωστρεφής είναι αυτή η συζήτηση και προσανατολισμένη στον εαυτό μας. Αυτή η τεράστια πίεση που ζούμε αυτόν τον καιρό και αισθανόμαστε προβλημάτων είναι τελικά το αποτέλεσμα μιας στρεβλής πολιτικής προσφύγων και μεταναστών έσω στρεφούς που ακολουθούσαμε επί δεκαετίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βολευτεί με το Δουβλίνο όλα αυτά τα χρόνια που είχε στόχο την περιχαράκωση και τον περιορισμό του προβλήματος στις παραμεθόριες χώρες. Και αν δεν μας είχε ταρακουνήσει αυτό που συμβαίνει, που βουλιάζουν τα σκάφη στη Μεσόγειο, είχαμε πέσει και σε μια αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Νότος της Μεσογείου. Δεν είναι απλή η κατάσταση τώρα να βγεις από ε, ε, αυτή την διάθεση αδιαφορίας, εφησυχασμού και περιχαράκωσης. Αλλά είναι αρκετά ισχυρή η Ευρώπη να τα καταφέρει αν σταματήσουμε να καταστρέφουμε και να κινδυνολογούμε ε, για την Ευρώπη σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Γιούνκερ, είναι σημαντικές οι αποφάσεις που ελήφθησαν για να γίνουν περισσότερα έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των προσφύγων στην Τουρκία και σε άλλες γειτονικέ χώρες της Σύριας. Αυτό όμως που θεωρώ σφάλμα, και είναι παλιό σφάλμα αυτό, είναι ότι για να κάνουμε κάτι σωστό, συμμαχούμε και πάλι με κάποιον ο οποίος κάνει λάθος πράγματα στη χώρα του. Μιλώ για τον πρόεδρο Ερντοάν. Αυτή τη στιγμή που συζητούμε εδώ, ένα μεγάλος ε, όμιλος τύπου, ε, πολιορκείται από την αστυνομία η οποία θα τον καταλάβει για να το διαχειρίζονται οι άνθρωποι του ΑΚΠ. Φανταστείτε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Ε, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε το Σαββατοκυριακό με τη Σύνοδο Κορυφής για τα Βαλκάνια και θεωρώ επίσης ρηξικέλευθο και καμπή αυτό που έγινε. Είναι ανθρωπιστική κρίση αυτό που ζούμε και ανθρωπιστική καταστροφή, όχι μόνο στην Ουγγαρία και στα Βαλκάνια. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να το λύσει αυτό. Να φροντίσει καλύτερα για τους ανθρώπους που ήρθαν σε εμά φεύγοντας για να βρουν καταφυγή και έφυγαν από τις χώρες τους που είναι κατεστραμμένες και βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα χώρο που θα προστατευτούν και εμείς έτσι λειτουργούμε υπέρ των πολιτών. Δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω ότι πιστεύω επίσης ότι εκτός από την οξία τώρα καταπολέμηση της ε, κατάστασης, θα πρέπει να σκεφτούμε και για μακροπρόθεσμες αλλαγές. Τι θα αντικαταστήσει τον κανονισμό του Δουβλίνου, τι θα γίνει μελλοντική προσφυγική πολιτική και μεταναστευτική πολιτική και πώς θα βάλουμε τάξη στα σύνορά μας και να βάλουμε τάξη όχι με περιχαράκωση, όχι με στρατιωτικοποίηση όπως εν μέρει κάνει η Frontex, αλλά με ευρωπαϊκές αξίες, με διεθνές δίκαιο, με ανθρώπινα δικαιώματα και με μια νέα στάση ανοιχτή και δίκαια και να ε, είμαστε γνώμονας για τη διαμόρφωση της νέας πολιτικής συνόρων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάρμς από την ομάδα του. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Φαράζ. Πρόεδρε, αυτή η κρίση των μεταναστών αρχίζει να καταλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι υπαρξιακή κρίση όντως. Ποια είναι η πραγματική φύση όμως των προτάσεων που έχουμε. Μιλήσαμε πολύ για δικαιώματα, ας πούμε και για τα δημοκρατικά τι αυτά. Υπάρχει μια αυταρχική Ευρωπαϊκή Ένωση που καταστρέφει τα δημοκρατικά δικαιώματα. Κάθε φορά που βλέπουμε κάποια κρίση χάνει η εθνική δημοκρατία. Το είδαμε το 11 ο Ιταλός Πρωθυπουργός ο τότε Μπερλουσκόνη. Απομακρύνθηκε και αντικαταστάθηκε από κάποιον αχυράνθρωπο. Στην Ελλάδα το 11 ο κύριος Παπανδρέου απείλησε δημοψήφισμα για το ευρώ και αντικαταστάθηκε πάλι από αχυράνθρωπο. Και σε αυτή την κρίση των προσφύγων λοιπόν, των μεταναστών μάλλον, βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες σαν την Ουγγαρία δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην μεταναστευτική πολιτική ούτε να αναγκαστούν να δεχτούν πράγματα που τα έχουν απορρίψει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας που καθόταν εκεί απέναντι είχε κερδίσει γενικές εκλογές και ήρθε για να του πούνε ότι είναι απαράδεκτα τα αποτελέσματα και πρέπει να αλλάξουν. Όλα αυτά όμως έφτασαν σε ένα καινούριο ναδύρ αυτή την εβδομάδα με την Πορτογαλία. Δεν το έγραψαν καθόλου τα μέσα. Μετά τις ε, γενικέ εκλογές μια αριστερή πλειοψηφία με σοσιαλιστικό σχέδιο είχε την πλειοψηφία και όμως ο πρόεδρος της Πορτογαλίας ο κύριος Σίλβα δεν τους δίνει την εντολή διότι λέει ότι αντιπροσωπεύουν αντιευρωπαϊκές δυνάμεις και επιτρέπει στη συντηρητική μειοψηφία να παραμείνει στην εξουσία. Αυτό, αυτό είναι η σύγχρονη εφαρμογή της, του δόγματος Μπρέσνιεφ. Ακριβώς αυτό γίνεται, γινότανε στις χώρες δορυφόρους της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό έγινε και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Μια χώρα έχει δημοκρατικά δικαιώματα μόνο αν είναι υπέρ του ευρωπαϊκού σχεδίου. Αλλιώς αφαιρούνται τα δημοκρατικά δικαιώματα, καταργούνται. Να μην μας εκπλήσουν όλα αυτά. Ο κύριος Γιούνκερ μα είπε και πριν ότι δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατική επιλογή κατά των ευρωπαϊκών συνθήκων. Και ο Γερμανός υπουργό Οικονομικών κύριο Σόιμπλε είπε οι εκλογέ δεν αλλάζουν τίποτα. Οποιοςδήποτε πιστεύει στη δημοκρατία βλέπει ότι η Πορτογαλία είναι η τελευταία τέτοια προσπάθεια με τελικό αποτέλεσμα να καταστραφούν, να καταργηθούν τα ατομικά δικαιώματα και τα εθνικά. Η χώρα μου ήταν πάντα υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και το διακινδύνευσε πολλές φορές για να προστατέψει την κοινοβουλευτική δημοκρατία όχι μόνο για τον εαυτό της αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και πιστεύω ότι όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία θα έπρεπε να ζητήσουν να επανειδρυθεί και το δημοψήφισμα στην Αγγλία δίνει μια τέτοια χρυσή ευκαιρία. Παρακαλώ. Κύριε Λαουριστίν. Ε, you compared situation Συγκρίνατε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Πορτογαλία με την πρώην ΕΣΤ. Ξέρω ότι δεν έχετε πείρα ζώντας υπό την πότα της ΕΣΤ. Εμείς έχουμε ζήσει. Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα όπου ο Μπρέσνεφ ή κάποιος άλλος αρχηγός αντιμετώπισε ελεύθερες εκλογές σε οποιαδήποτε πρώην δημοκρατία της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ήμουν παρόν τότε στην Ουγγρική εξέγερση, αλλά το έχω μάθει. Ξέρω τι έγινε και το 68 στην Τσεχοσλοβακία. Να σας πω τι λέει το δόγμα το το Όταν δυνάμεις εχθρικές προς τον σοσιαλισμό αναπτύσσονται σε μια σοσιαλιστική χώρα προς την κατεύθυνση του καπιταλισμού, τότε αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της χώρας αυτής, αλλά κοινό πρόβλημα και που ενδιαφέρει όλες τις σοσιαλιστικές χώρες. Πρέπει λοιπόν να αλλάξετε τη λέξη σοσιαλισμό με Ευρωπαϊστική Ένωση και θα δείτε τι αποτέλεσμα βγαίνει. Τώρα, από την ομάδα ΕΝΕΦ το λόγο έχει ο κύριος Δεκράφ. Πρόεδρε, η κυρία Μέρκελ την περασμένη εβδομάδα πήγε στο Σουλτάνο της Τουρκίας, η καγκελάριο της Ευρώπης, και συμφώνησαν ε, να μπει γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ένωση με αντάλλαγμα ε, την προσφυγική κρίση. Η δημοκρατία έχει πεθάνει. Η Γερμανία αποφασίζει για όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοκαταργείται και δημιουργείται μια νέα Οθωμανική αυτοκρατορία. Τα εξωτερικά σύνορα μας δεν είναι ασφαλή, ε, αλλά τα εσωτερικά σύνορα έχουν πέσει. Η ευρωπαϊκή ελίτ που κάθεται εκεί ε, προσανατολίζεται στο θηρίο της Άγκυρας και παραδίδεται. Δεν ισχύουν πια τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεργάζεται με το Ισλαμικό κράτος ο Ερτογάν, βομβαρδίζει τον πληθυσμό του. Ε, όλα αυτά δεν μας απασχολούν. Μόνο στο 1913 εκδιώχθηκαν ε, από τα Βαλκάνια οι Τούρκοι και σταμάτησαν να διώκουν τους χριστιανούς. Και τώρα θέλουν να ξαναγυρίσουν στην Ευρώπη. Όπου υπάρχει το Ισλάμ, η γυναίκα είναι δεύτερης κατηγορίας, τα ε, παιδιά πουλιούνται σε σκλαβοπάζαρα και κυριεύουν παντού ε, η βία και η κυρία ε, Μέρκελ υπερασπίζεται ε, χριστιανικές αξίες και αξίες της Δύσης, τις οποίες τώρα απεμπολεί. Έχουμε βιαιότητες κατά των χριστιανών, βιασμούς σε πολύ μεγάλη κλίμακα και αυτό θα γίνει σε κάθε κράτος, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό. Αυτό εστί το Ισλάμ. Ε, θέλουν να κατακτήσουν τη Δύση και να την καταργήσουν. Σταματήστε αυτή την επέλαση, κλείστε τα σύνορα και μην αφήσετε ποτέ την Τουρκία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τους μη εγγεγραμμένους, το λόγο έχει τώρα η κυρία Ντότς. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ακούγοντας τη σημερινή συζήτηση, ελπίζω όσα ακούσαμε να είναι μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση σε αυτά που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες με τους πρόσφυγες και μετανάστες που βαίνουν προς την Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από αυτούς φεύγουν από την καταδίωξη και από τον πόλεμο, αλλά δυστυχώς ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη βοήθησαν τους ε, διακινητές έτσι ώστε να μειώσουν τους πιο ευάλωτους. Ε, κύριε Τούσκ, σήμερα μιλήσατε για την προστασία των συνόρων, γιατί καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να μας υποκαταστήσει στην ε, υπεράσπιση των συνόρων μας. Κύριε Γιούνκερ, Είπατε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ανεξέλεγκτο αυτό ρεύμα μετανάστευσης. Αυτό είναι μέρος όμως της απάντησης. Χρειάζεται διτή απάντηση, σταθερότητα στην περιοχή και ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Όμως με ενοχλεί η στάση πολιτικών αρχηγών. Κύριε Βέμπερ, ε, στην ουσία προβήκατε σε μία έκρηξη και αυτό ε, έναντι ημών. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι των άκρων. Εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους Σύριους έμπρακτα και είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος ε, διμερής δωρητής βοήθειας προς τη Σύρια και μία από τις λίγες χώρες που ανταποκρίνεται στους στόχους της χιλιετίας είναι πονίδιστο γιατί από τους Προέδρους Συμβουλίου και Κομισιόν, ενώ ακούσαμε πολλά για τις ευρωπαϊκές χώρες και χρηματοδότησή τους, αγνοήσατε την ε, ε, βοήθεια των χωρών του Περσικού κόλπου, την ενδυνάμει αυτή η βοήθεια. Θα πρέπει αυτές οι χώρες να αναλάβουν την ηθική τους ευθύνη για να αντιμετωπίσουν την κρίση όπως και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Το λόγο τώρα έχει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κύριο Ροέλ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τεράστιο πρόβλημα το ζήτημα των προσφύγων και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα είναι ότι από πρωί ως το βράδυ ακούω όλους να περιγράφουν την κατάσταση πόσο δύσκολη είναι και πόσο περίπλοκη. Άλλοι λένε ποιο στέει και τι πρέπει να γίνει. Ο τρίτος λέει τι έγινε λάθος στο παρελθόν. Συνεδριάζει το Συμβούλιο και μετά από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει αποφάσεις για συγκεκριμένα μέτρα και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό εκνευρίζει τον κόσμο. Εμείς ως πολιτικοί έχουμε ως δουλειά όχι να συζητούμε τα προβλήματα και να τα αναλύουμε, ούτε να αλληλοϊβριζόμαστε, αλλά να τα λύνουμε. Ο κόσμος αντιμετωπίζει διαφορετικά το προσφυγικό όταν βλέπει ότι λειτουργεί η πολιτική και κάνουν οι πολιτικοί αυτά για τα οποία δεσμεύονται. Δεν είναι φυσιολογικό να εφαρμόσεις αυτά που έχεις αποφασίσει και έχεις συμφωνήσει. Έχουμε πολλά προβλήματα στην Ευρώπη που δεν θα τα είχαμε αν τηρούσαμε ο καθένα στα συμφωνηθέντα, στα εκάστοτε όργανα. Και δεν χρειάζεται κάθε φορά να τα ξανανοίγουμε. Πάει αυτό. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που διοργανώσατε αυτό τη σύνοδο το Σαββατοκύριακο. Είπατε να καθίσουμε με του ενδιαφερόμενου, να ανταλλάξουμε και να ορίσουμε ποιο θα κάνει τι. Και βέβαια δεν είχαν όλοι παρόντε. Και βέβαια δεν ήταν κάποια τυχαία συνεδρίαση ε, και βέβαια δεν είναι όλες οι αποφάσεις το απάβγασμα της σοφίας αλλά είναι επιτέλους κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ορίστηκαν, αποφασίστηκαν για να βοηθήσουν κόσμο και να λύσουν προβλήματα και έχω μια πολύ απλή προσδοκία όλοι οι συμμετέχοντες, είτε είναι η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Συμβούλιο που έχει την πιο πολλή δουλειά εδώ, να κάνουν αυτό για το οποίο δεσμεύτηκαν το χέρι στην τσέπη, να δώσουν λεφτά στην Κομισιόν με δυνατότητες να δράσει και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Frontex να μπορέσει να λειτουργήσει, να είναι αποτελεσματική, με στελεχωμένη. Ε, αν δεν μπορούν μόνα τους τα κράτη-μέλη, έχουμε εργαλεία, ας το χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν ένα πρώτο βήμα και ως πρώτο θα ακολουθήσει και δεύτερο φυσικά και γι' αυτό ήταν σωστό. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω καταρχήν, πριν δώσω το λόγο στην ε, κυρία Φαγιόν, θα ήθελα να κάνω μία έκκληση. Σας παρακαλώ να αρκεστείτε στο χρόνο σας. Ήδη έχουμε αργήσει. Θα γίνει η ψηφοφορία και τότε ε, ο κύριος Τούσκ και ο κύριος Γιούνκερ θα πρέπει να μιλήσουν, πριν δηλαδή από την ψηφοφορία. Ήδη η ψηφοφορία είναι δύσκολη και στις 3 ε, η ώρα έχουμε άλλη συζήτηση. Σας παρακαλώ να ε, παραμείνετε στο χρόνο σας και να μην τον υπερβαίνετε. Η κυρία Φαγιών έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ήδη επισκέφτηκα ένα κέντρο καταβλισμού στα ε, σύνορα της Σλοβενίας. Είδα πολλά κουρασμένα, αδύναμα ε, πρόσωπα. Τι γίνεται όμως με την ε, Κροατία. Η Κροατία δεν θα πρέπει να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα τη στιγμή που πρέπει να εγκαταστήσει και άλλες σκηνές όπως έκανε χτες. Όταν ε, μιλώ στους Σλοβένους πολίτες, βλέπω ότι στην ουσία υποβαθμίζουμε την αξιοπιστία μας, διότι αποστέλουμε τους πρόσφυγες από το ένα σημείο στο άλλο. 80.000 πρόσφυγες μπήκαν στη Σλοβενία τις τελευταίες ε, μέρες. Είναι σαν να έμπαιναν 3.200.000 στη Γερμανία. Δυστυχώς η Σλοβενία έχει γονατίσει, θα επικρατήσει χάος και πιστεύω ότι οι ξενόφοβοι θα βγουν αληθινοί. Δεν λέω ότι δεν μπορούν να γίνουν πράγματα επί της ουσίας, αλλά θα πρέπει να ε, λάβουμε αποφάσεις με βάση το τι μας λέει η καρδιά μας, Λεγκούτκο, για δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, οι αριθμοί έχουν σημασία αλλά δεν κολλάνε. Φέτος 700.000 μετανάστες ήρθαν στην Ευρώπη αλλά μας λένε επίσης ότι 800.000 άνθρωποι ήρθαν στη Γερμανία ότι κάθε μέρα 5.000 άνθρωποι περνάνε τα σύνορα και στις βαλκανικές χώρες και στις μεσογειακές χώρες και δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολύ δυνατός στα μαθηματικά για να καταλαβαίνει ότι ο πρώτος αριθμός 700.000 είναι λάθος. Είναι ψηλότερος ο αληθινός αριθμός. Εδώ μέσα ακούστηκε ότι τα επόμενα χρόνια περίπου 16 εκατομμύρια άνθρωποι μάλλον θα φύγουν από τις χώρες τους στις ταραγμένες περιοχές ψάχνοντας ένα καλύτερο μέλλον αλλού και ο πρόεδρος Τούσκ είπε ότι αυτά που βλέπουμε τώρα μπορούν να συγκριθούν με τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές των, της προϊστορικής εποχής. Αν τουλάχιστον ένα τρίτο από αυτά τα 16 εκατομμύρια έρθει στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε ένα καινούριο μεσαίο μεγέθους έθνος στην επικράτειά μας. Τι σημαίνουν οι αριθμοί αυτοί. Πρώτον, οι πολιτικοί κρύβουν τους πραγματικούς αριθμούς. Δεύτερον, τα εργαλεία που προτείνει η Ένωση δεν αρκούν. Και τρίτον, έχω το αίσθημα ότι αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται μάλλον για να επιβληθεί η ισχύ της Ένωσης πάνω στα, κράτη, στα έθνη κράτη παρά για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η στρατηγική λοιπόν αυτή είναι αποτυχημένη, αλλά το μέλλον μπορεί να είναι ακόμη χειρότερο. Ο κύριος Ντεπρέ, για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επίτροπης για την πρωτοβουλία που έλαβε και τα μέτρα που ενέκρινε τα 17 μέτρα. Είδαμε αυτές τις τρομακτικές εικόνες προσφύγων που έπρεπε να διαβούν έναν ε, παγωμένο ποταμό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Τα εξωτερικά σύνορα είναι κοινά σύνορα. Αυτό το υπενθυμίσατε. Και αυτό που είναι κοινό θα πρέπει να το διαχειριστούμε ως κοινό. Μην μου πείτε ότι η Frontex έχει τα μέσα που θα έπρεπε. Η Frontex στην ουσία είναι ένας ζητιάνος που ζητά από τα κράτη-μέλη ε, εξοπλισμό, βοήθεια της ακτοφυλακής, συνοριοφύλακες και ούτω καθεξής. Εάν θα πρέπει να διαχειριστούμε τα κοινά σύνορα θα πρέπει να ξαναδούμε το καθεστώς της ε, Frontex, η οποία να ακολουθεί τους ε, κοινούς ε, ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς και μέτρα. Μιλήσατε για συνεργασία με τις χώρες διέλευσης, όπως την Τουρκία, αλλά να διαπραγματευτούμε με τον Ερντογάν, ο οποίος στην ουσία λέει ότι αντιμετωπίζει τους ε, τρομοκράτες, αλλά δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βοηθά τους ε, διακινητές, ιδιαίτερα στο Μποντρούμ. Γιατί για μια συγκυριακή βοήθεια το αντιστάθμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει παρά να είναι συγκυριακό και όχι διαρθρωτικό και μόνο. Η κυρία Αλμπιόλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ η Σλοβενική αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα στους πρόσφυγες, άνδρες και γυναίκες. Σλοβενία, φιλελεύθερη κυβέρνηση, Ουγγαρία, κυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, χρησιμοποιεί σκυλιά, αντλίες νερού και δακρυγόνα στα σύνορα και στους καταβλισμούς, 16 Οκτωβρίου. Βουλγαρική αστυνομία πυροβολεί και σκοτώνει έναν Αφγανό στα σύνορα, Βουλγαρία, ε, κυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αλλά αυτό που σίγουρα ε, καθορίζει και ορίζει καλύτερα ε, τη σχέση μας είναι η κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας που τους βάζει αριθμούς στα χέρια και η Γερμανία έχει ανοίξει τον Ταχάου και το έχει κάνει καταβλισμό, το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, μηδέν από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από το Φιλελεύθερο Κόμμα διώχνουν τους συναδέλφους από την Ουγγαρία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία μηδέν. Κυρώσεις της Ένωσης προς χώρες αυτές μηδέν. Κύριε Γιούγκερ, κύριε Πιτέλα, κύριε Βέμπερ. Τα δικά σας κόμματα, οι δικές σας κυβερνήσεις ε, ε, δεν επιδεικνύουν αλληλεγγύη αλλά παραβιάζουν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Κέλλερ, για ένα λεπτό. Excuse me. Ο πρόεδρος. Υπάρχει μία μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Go on. Ναι, παρακαλώ. Πέτερλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να αντιδράσω οπωσδήποτε σε αυτή αυτή την ε, αντίδραση συναδέλφου για τη Σλοβενία και τον τρόπο της. Πώς θα αντιδρούσατε εσείς όταν, αν υπήρχε μία ε, κατάσταση σύραξης μεταξύ των ίδιων των μεταναστών. Θεωρώ ότι οι Σλοβαίνοι έδρασαν με μεγάλη υπευθυνότητα. Νομίζω ότι υπεύθυνη δράση σημαίνει να σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί δακρυγόνα απέναντι σε ανθρώπου που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βαρβαρότητα και τον πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι τρόπο αυτό. Η κυρία Κέλλερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ περίεργος πώς δεν απογοητεύομαι τόσο πολύ ε, από όσα προέκυψαν από την Κυριακή, όπως είπαν ο κύριος Σόλτς και κάποιοι άλλοι. Ε, διαφωνώ, γιατί επιτέλους ε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατάφεραν να καταλάβουν ότι είναι ανθρωπιστική η κρίση. Βεβαίως οι πρόσφυγες θέλουν τροφή, στέγη, νερό, αυτά που είπατε κύριε Γιούνκερ, αλλά επιτέλους για αλλαγή το έχουμε και στα συμπεράσματα. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν και πραγματικότητα όλα αυτά. Και επίσης χαίρομαι που η Σύμβαση Γενέβης και το κοινοτικό δίκαιο τονίστηκε, δεν ξέρω πώς αυτό θα συγκεραστεί με τις επαναπροωθήσεις στο Αφγανιστάν, διότι οι Αφγανοί πρόσφυγες έχουν αναγνωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόσφυγες και σχεδόν ε, είναι στο κατόφλι του 75% για να είναι επιλέξιμη για επανακατάσταση. Άρα φυσικά το Αφγανιστάν δεν είναι ασφαλής χώρα και δυστυχώς την Κυριακή η Μήνη Σύνοδος δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα ζητήματα ε, της δίκαιης κατανομής δίκαιης και για τα κράτη και για τους πρόσφυγες και για τη ε, νόμιμη πρόσβαση. Αυτό θα πρέπει εμείς να κάνουμε. κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μερικές παρατηρήσεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής. Πρώτον, επιτέλους παραδεχθήκαμε ότι η Ευρώπη δεν ε, προστατεύει μέχρι τώρα ε, σωστά τα εξωτερικά της σύνορα. Αποφασίστηκαν κάποια μέτρα, είναι θετικά καταρχήν. Δεύτερο, 10 δισεκατομμύρια θα δώσει το Συμβούλιο για τις χώρες Αφρικής και Ασίας με την ελπίδα να σταματήσει αυτό τις μεταναστευτικές ροές, ε, οποία αφέλεια. Και τρίτον, ε, συνάδελφοι, χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική μετανάστευσης που να λέγει ότι η Ευρώπη ανοίγει τα σύνορά της μόνο για πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές. Τελεία. Και αποφάσεις που λαμβάνονται ε, θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε ό,τι αφορά ε, την υποδοχή των προσφύγων από διάφορες κυβερνήσεις και χώρες δεν θα πρέπει να αντιδρούμε και να παρουσιάζουμε την κατάσταση διαφορετική στρεβλώνοντάς τη. Ο κύριος Μπριουά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Διαδέχονται οι σύνοδοι στην Ευρώπη μια την άλλη και διευρύνονται ε, οι ροές. Η δήμαρχος του Καλέ, του Ι.Μ.Π. είπε πρώτα ότι είναι οι παράνομοι ε, μετανάστες ε, πολιτιστικός πλούτος και τώρα ζητούν από κάποιους πολίτες να μεταναστεύσουν οι ίδιοι και να αποδημήσουν πλήρης αναρχία και φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπόδουλες κυβερνήσεις που αρνούνται να ανακτήσουν τον έλεγχο των συνόρων τους. Γι' αυτό η σύνοδος της Βαλέτας δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα, διότι επιμένει και παραθέτω στην προώθηση των νόμιμων οδών μετανάστευσης και την ενίσχυση της προστασίας των μεταναστών. Ε, αντίστροφα με αυτές λοιπόν τις ανεύθυνες ε, θέσεις ζητώ την πλήρη αναστολή και διακοπή των συμφωνιών Σέγγεν και την ενίσχυση των ελέγχων στα εθνικά σύνορα έτσι ώστε οι μετανάστες να κρατούνται σε κέντρα κράτησης και να απελάβνονται αμελητοί στις χώρες ε, καταγωγής τους. Ιδού λοιπόν το σαφές μήνυμα στους μετανάστες να μην μας κουβαλιώνται εδώ. Κύριος Σαπιτίδιος, για ένα λεπτό. Οι αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 15 Οκτωβρίου είναι αποτέλεσμα του πανικού που έχει καταλάβει τους ηγέτες των χωρών της Ευρώπης από την αθρώα και ξαφνική εισβολή χιλιάδων παρανόμων μεταναστών και τις ανικανότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν την κρίση που προέκυψε από το πρόβλημα αυτό έτσι το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να αναβαθμίσουν το ρόλο της τουρκίας μιας χώρας η οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και για τη δημιουργία αλλά και για την όξυνση του μεταναστευτικού προβλήματος. αντί η ευρωπαϊκή ένωση να απαιτήσει από την τουρκία η οποία σημειωτέων και ότι δεν πληρεί τα κριτήρια της συνθήκης της κοπενχάγης είναι προς ένταξη χώρα να εκπληρεί τις υποχρεώσεις της και να μην προωθεί χιλιάδες παρανόμων μεταναστών στην ελλάδα την ανέχεται να εκβιάζει την κύπρο με διχοτόμηση αν δεν υποκύψει στις πιέσεις και τις απαιτήσεις της και παράλληλα διαστόματος της κυρίας Μέλκερ προσφέρει 3 δισεκατομμύρια ε, ευρώ στον κύριο ερντογκάν παρά το γεγονός ότι αυτός αρνείται να τα λάβει και θέλει περισσότερα και ενδεχομένως διπλάσια. πιέζει την ελλάδα να έχει κοινή συνεργασία εκτοφυλακή της με την τουρκική. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που έχει σημασία είναι... Αυτό που έχει σημασία είναι να σας πω ότι δέχομαι απόλυτα τη διάγνωση του κυρίου Τούσκ. Η μετανάστευση έχει αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική σκηνή σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Εάν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο αριθμός των προσφύγων είναι σωστός, θα πρέπει να δούμε ότι αποτελούν πραγματική και ουσιαστική πρόκληση για όλα τα κράτη μας και έχει μεγάλη σημασία γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες στις χώρες της Μέσης Ανατολής και στην Αφρική, δηλαδή ε, από εκεί που προέρχεται το πρόβλημα. Συμφωνήσαμε ότι οι προτεραιότητες μας θα είναι να προασπίσουμε τα σύνορά μας και ε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν είναι τόσο διάτρητα τα σύνορά μας, διότι αυτό οδηγεί στις ροές που έρχονται ιδιαίτερα από τη Συρία, στην προσέλκυση δηλαδή αυτών των ροών. Συμφωνήσαμε με βοήθεια ενός δις για τους πρόσφυγες της Μέσης Ανατολής. Αρκεί αυτό. Μάλλον όχι. Πρέπει να βοηθήσουμε και την ε, Τουρκία. Έχει 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες πλέον η Τουρκία. Ίσως η Τουρκία θα μπορούσε να σταματήσει αυτή τη μεγάλη πίεση που βρίσκεται ενώπιον των πυλών μας. Θα θέλαμε να βελτιωθεί η κατάσταση στη Συρία, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και να συνεργαστούμε και με τα Ηνωμένα Έθνη για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή κρίση. Έχετε μπλε κάρτα. Τη δέχεστε. Έχουμε ή δεν έχουμε. Ναι, εντάξει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Δεν αναφερθήκατε σε αριθμητικά στοιχεία, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω έχετε πραγματικά ουσιαστικά αριθμητικά στοιχεία και αναλογίες ως προς τους ε, πρόσφυγες, ποιοι είναι επιλέξιμοι για χορήγηση ασύλου και πόσοι θα πρέπει να επιστρέψουν. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ συνάδελφε, δεν ε, έκανα κατανομή ε, ως προς τους οικονομικούς μετανάστες και τους πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κατανομή τώρα. Χρειάζεται μία εις βάθος ανάλυση. Αν είχαμε ένα σωστό σύστημα καταγραφής θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι 700.000 μέχρι το Σεπτέμβρη μπήκαν στα σύνορά μας, αλλά θα πρέπει να γίνει εις βάθος ανάλυση και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπαν ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων για να δούμε ποιοι είναι οι ε, οικονομικοί μετανάστες και ποιοι όχι. Φλέκενστάιν, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να επανέλθω στη Σύνοδο Κορυφής ε, είναι πραγματικά θλιβερό αρκετά ε, να δούμε τι χαρακτηρίζουμε ως επιτυχία. Θέλω να υποστηρίξω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Τίμερμανς να κάνετε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Ε, το αξίζουν διότι έχουν τόσο καιρό εκεί τους Σύρους πρόσφυγες και δεύτερον μας δίνει ένα περιθώριο να ανασάνουμε λίγο, να δημιουργήσουμε τις υποδομές για να μπορούμε να τους υποδεχόμαστε καλύτερα τους ανθρώπους αυτούς που είναι πρόσφυγες και εκείνους που τους καλωσορίζουν. Αλλά δεν θα πρέπει να απεμπολίσουμε τις αξίες και τις αχαίριμες μας. Δεν το πιστεύει κανείς ότι γίνεται κάτι τέτοιο στις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν μπορούμε να το λύσουμε με την ηθική και μόνο. Δεύτερον, Προσπαθήστε να κάνετε ό,τι μπορείτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, τη Ρωσία, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Συρία. Μόνο από κοινού θα μπορέσουμε να το λύσουμε και χωρίς ρεαλισμό δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Γιούγκερ, μέσα σε πέντε μέρες την περασμένη εβδομάδα και παρά τη θαλασσοταραχή τα νησιά του αιγαίου πλημμύρισαν από 48.000 νέους πρόσφυγες που ήρθαν να προσθεθούν στους 450.000 πρόσφυγες που είχαν ήδη κατακλείσει την Ελλάδα από τις αρχές του χρόνου. Με βάση τη ρήτρα κατανομής προσφύγων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την έκταση, τον πληθυσμό και το ΑΕΠ κάθε χώρας που αποφάσισε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ελλάδα πρέπει να φιλοξενήσει το πολύ 11.000 πρόσφυγες. Και όμως με εργαλείο το μνημόνιο, στην προχθεσινή μίνι σύνοδο των Βρυξελών, ουσιαστικά επιβλήθηκε στην ελλάδα να φιλοξενήσει πενταπλάσιο αριθμό προσφύγων που θα φτάσουν τις. πενήντα χιλιάδες κύριε juncker η ελλάδα δεν μπορεί να μετατραπεί σε μια τεράστια φαβέλα προσφύγων. ο φτωχοποιημένος από τα μνημόνια ελληνικός λαός δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους πρόσφυγες και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. όπως επίσης κύριε juncker πρέπει να καταλάβετε ότι η φύλαξη των ελληνικών σύνορων ανήκει στα κυριαρχικά δικαιώματα της ελλάδας. κύριε juncker ήρθε η ώρα να πάψετε να θοπεύετε την τουρκία και να την αναγκάσετε να βάλει τέλος στα δουλεμπορικά κυκλώματα που λειτουργούν στην επικράτειά της. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί ε, οργανώσατε αυτή την ε, συνάντηση την Κυριακή για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Δεν δέχομαι την επικριτική σας στάση εναντί των αρχηγών των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που υπερβαίνει τις δυνατότητές μας κατά 100%. Όμως η συνάντηση ήταν χρήσιμη. Η Σλοβενία είναι μια μικρή χώρα, βρίσκεται στο μονοπάτι των Δυτικών Βαλκανίων και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν αποτελεί φυσική καταστροφή, αλλά είναι απότοκο καταστροφικών αποφάσεων που έλαβαν πολιτικοί. Οι μεγάλες μάζες προσφύγων ήρθαν σε μας, βρίσκονται ενώπιον των πυλών μας, όπως και στο παρελθόν και το δεχόμαστε αυτό. Δεχτήκαμε ανθρώπους από διάφορες θρησκείες, αλλά σήμερα είμαστε διαφορετικοί. Θα πρέπει να δράσουμε με βάση τις αξίες μας. Αυτό αφορά τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ και θα πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές λύσεις αποφεύγοντας τη μυσαλλοδοξία. Κύριος Παπαδεμόλης, για ένα λεπτό. Ναι. Κύριοι της Κομισιόν και κυρίως του Συμβουλίου, είναι η ώρα από τα λόγια να περάσετε στα έργα και μέχρι τώρα έχουμε καθυστέρηση και αναβολή ακόμη και στην υλοποίηση αποφάσεων που έχετε πάρει. χρειάζεται μια βιώσιμη ευρωπαϊκή λύση ανθρωπιστική στο πρόβλημα των προσφυγικών ροών. αν αυτή δεν δοθεί κινδυνεύει με μια διαλυτική κρίση η ίδια η ευρωπαϊκή ενοποίηση και απειλείται η ευρώπη με την αναβίωση και την ενίσχυση ξενοφοβικών ρατσιστικών φασιστικών απόψεων. η χώρα μου η ελλάδα δεν αντέχει να σηκώνει μόνη της το βάρος και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών. και έρχεται χειμώνας και το αιγαίο κάθε μέρα γίνεται νεκροταφείο. πότε θα αλλάξει επιτέλους το δουβλίνο 2. πότε θα πάρετε ειρηνευτικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Συρία. Πότε επιτέλους θα εφαρμόσετε με ελαστικότητα το σύμφωνο σταθερότητας στις χώρες που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και είναι πολύ θετικό και το λέω και προς εσά, κύριε Γιόνκερ, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνέβη καν αυτή η συνάντηση την Κυριακή. Γιατί ακριβώς εκεί έγκυται το μέλλον της Ευρώπης. Να καθόμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι και όχι ο ένας να ορθώνει τύχη απέναντι στον άλλον και ακαθωτά σειρματοπλέγματα. Σε ένα κοινό τραπέζι να συζητάμε για μια κοινή λύση. Και είπατε κι εσείς ο ίδιος αυτό θα πρέπει να είναι η φυσιολογική κατάσταση. Δυστυχώς δεν είναι ακόμα. Χρειάζεται υποστήριξη και για χώρες που δεν είναι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι χώρες των Βαλκανίων. Πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Τώρα έρχεται και χειμώνα. Είναι πρόσφυγες οι άνθρωποι που φεύγουν από βόμβες και από πόλεμο να γλιτώσουν. Κάτι άλλο που λείπει και φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι αυτά που έχουν τάξει τώρα τα κράτη-μέλη πρέπει να τα εφαρμόσουν. Χρειάζονται χρήματα αλλά και δίκαιη κατανομή των προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη. Στο χέρι σα, είναι κύριε Τούσκ τώρα να πιέσετε επιτέλου, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου να πιέσετε τα κράτη-μέλη και να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Ένα κοινό σύστημα ασύλου θα ήταν αυτό που χρειάζεται και χρειάζεται τώρα για να μην τσακωνόμαστε και να μην στρεφόμαστε ο ένα κατά το άλλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καστάλντο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Ενώ, ενώ ε, η Ρώμη καίγεται, εμείς ε, με Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συζητήσεις που έγιναν και μέσα στα πλαίσια του Σέγγεν. Αυτές οι ροές της απόγνωσης ε, βρίσκονται στις χώρες μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε 260.000 ε, ανθρώπους που πρέπει να περάσουν από την Κροατία και μόνο. Μιλάμε όμως για μία Frontex και για την αντιμετώπιση των διακινητών. Ε, έχουμε να κάνουμε με μία δαμόκλειο σπάθη. Πώς όμως θα αντιμετωπίσουμε επί της ουσίας το ζήτημα. Πότε θα αρχίσει, θα γίνει αυτή η επανακατανομή. Πότε θα αναθεωρηθεί το Δουβλίνο ιδιαίτερα ως προς τις ε, πολιτικές μας ε, στην Συρία. Μία γραμμή έχουμε γράψει μόνο για να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της ε, κακοδεμανίας. Δεν ξέρουμε τι προσπάθειες καταβάλλονται. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να χαιρετίζουμε τον Ερντογάν σαν καλύτερο μας φίλο. Ενώ στην ουσία, όπως είπε ο Βερχόφστατ, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα διαγωνισμό υπάρχει ένα ενιαίο κόμμα που είναι το κόμμα του πολέμου. Αυτό επικρατεί και ενώ μιλάμε για την Μεσόγειο στην ουσία καίγεται ολόκληρη η Αφρική. Να πάρουμε νόμπελ υποκρισίας λέγω ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Άνεμανς, αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι πού θα φτάσει ο κινησμός ο κύριος ε, Γιούνκερ συγχαίρει την κυρία Μέρκελ που αγνοεί τις ε, δημοσκοπήσεις ε, του λαού για την πολιτική μετανάστευση. Δεν θα τα καταφέρουμε φαίνεται να λέει ο κόσμος, αλλά εμείς το αγνοούμε και το περιφρονούμε. Είναι μακράν η χειρότερη ε, ε, κατάσταση και η χειρότερη απόδειξη για τους πολίτες ότι δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες και τι πιστεύουν. Καμία σχέση με τη δημοκρατία. Ελεύθερη κυκλοφορία για αγαθά και πολίτες για να οργανώσετε τώρα τη μεταναστευτική κρίση, τη μεγαλύτερη της ιστορίας και οικονομικά και κοινωνικά φάνηκε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντικαταστήσει τους πολίτες της Ευρώπης. Κοιτάξτε το πραξικόπημα που έκανε στην Πορτογαλία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς έχει καταρρεύσει η δημοκρατία στην Ευρώπη. Πραγματικά είναι τρελή η πολιτική σας εκφιασμός και χειραγώγηση για τη μετανάστευση. Ε, είστε παρακαλώ ο, κύριε, ο χειρότερος προπαγανδιστής. Ο κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό παρακαλώ. είναι πολύ επικίνδυνες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους λαούς συνολικά η αποφάσεις της συνόδου πάει πολύ η ελληνική κυβέρνηση να προσποιείται ότι τάχα τις απέτρεψε γιατί η ελλάδα με αυτές μετατρέπεται σε σταθμός καταναγκαστικής συγκέντρωσης ε, σε καταβλισμούς πάνω από πενήντα εγκλωβισμένων προσφύγων σε μια νέα εκδοχή του δουβλίνου τα δε κέντρα διαλογής θα αποδέχονται τους πρόσφυγες με προσόντα κατά παραγγελία των μονοπωλίων και οι υπόλοιποι οι περισσότεροι θα ανακατευθύνονται πολύ απλά δηλαδή θα απελάβνονται πίσω στην κόλαση των πολέμων για τους οποίους ευθύνεται η ευρωπαϊκή ένωση οι ηνωμένες πολιτείες και το νατο. τα περί κοινών περιπολιών ελλάδας και τουρκίας μεθοδεύουν τη συνδιαχείριση στο αιγαίο ενώ η ανάθεση στο frontex ρόλου καταστολή σε πρόσφυγες στα ελληνοσκοπιανά και ελληνοαλβανικά σύνορα ε, και με συγκέντρωση δυνάμεων ταχεία επέμβαση σημαίνει να φυλά ο λύκος τα πρόβατα δηλαδή η ευρωπαϊκή ένωση τα σύνορα καταργώντα κάθε έννοια κυριαρχικού δικαιώματο. οι λαοί μπορεί να διεκδικήσουν άμεσα μέτρα στήριξη των προσφύγων και να αντιπαλέψουν τι υπεριαλιστικέ επεμβάσει του ευρωνοσιακού κανονισμού και μηχανισμού καταστολή σημαδεύοντα το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που γεννά πολέμου φτώχεια και προσφυγιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φτάνει πια. Η αδυναμία μας, οι αντιφάσεις μας, η υποκρισία μας φτάνει. Να πάρουμε τα μαθήματα που επιβάλλεται να πάρουμε από την έξοδο των μεταναστών. Πρώτον, η Ένωση δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει καταστάσεις κρίσης. Είναι θέμα διακυβέρνησης να αντιμετωπίσουμε μέχρι το 2040 την υπερθέρμανση του πλανήτη το ξέρουμε αλλά να συνοδεύσουμε και να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες δεν το ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Αντιδρούμε χαοτικά σε μια χαοτική κρίση. Δεύτερο μάθημα, τα χρηματικά. 100 δισεκατομμύρια λέει δολάρια για να μειώσουμε την υπερθέρμανση, α, πρωταθλητές ενώ να βοηθήσουμε ορισμένες εκατοντάδες ανθρώπους στα σύνορα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα μέσα. Σε λίγες μέρες θα εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του 16 τελείως ανεπαρκή. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να δεχτούν πρόσφυγες, αλλά κανείς δεν θέλει να πληρώσει ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι φτωχοί, ούτε οι μεγάλοι, ούτε Και τρίτο μάθημα, η πολιτική υποκρισία σε όλες μας τις χώρες, σε όλα τα επίπεδα και σχεδόν σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Άλλοι μιλάνε για αξίες, άλλοι μιλάνε για ιουδαιοχριστιανικές ρίζες, άλλοι για το διαφωτισμό, άλλοι για την ε, ένωση των προλεταρίων σε όλες τις χώρες. Και όλοι αναφέρονται στην παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά μέσα μπροστά στις κάλπες αυτοί που μιλάνε για τις καθολικές αυτές αξίες αφήνουν αδιάφορους τις γυναίκες, τα παιδιά που υποφέρουν διότι δεν είναι σαν και εμάς γιατί προέρχονται από αλλού. Καιρός είναι λοιπόν να διορθωθούν πνευματικά τα πράγματα αυτά και στην Ευρώπη και ευχαριστούμε κύριε Γιούνκερ που μας το υπενθυμίσατε. Δύο συνάδελφοι έχουν προβάλει μπλε κάρτα. Θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω και τους δύο να κατανοήσετε την κατάσταση και να συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Ε, Φρουνζουλίκα και Μπρετών, δέχεστε να μην υποβάλλετε ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυρία Σίπελ για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εθελοντική ένωση, αλλά τα κράτη-μέλη της υποχρεώνονται και αναλαμβάνουν συγκυριαρχία και κοινή ευθύνη. Τα παλιά και νέα κράτη-μέλη όμως και πάλι τείνουν να το λησμονούν αυτό και ε, πέφτουν σε εθνικούς εγωισμούς. Ε, βελτιωμένος έλεγχος στα σύνορα. Τι σημαίνει, θα πρέπει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πρόσφυγες να έχουν δυνατότητα νόμιμης πρόσβασης και ε, με ατομικές αιτήσεις ασύλου. Τώρα ε, η καταγραφή των προσφύγων και τα όσα προτείνονται μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον σύντομα γίνει η κατανομή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οργανωθεί η ένταξή τους και ταυτόχρονα βελτιώσουμε και την κατάσταση των προσφύγων σε άλλες χώρες. Κατά τα άλλα, η φορολογική δικαιοσύνη θα ήταν επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ένα θέμα αρχής που πρέπει να μας απασχολήσει. Οι εθνικοί εγωισμοί δεν αποτελούν λύση. Τα κράτη-μέλη τώρα θα πρέπει να δράσουν ως αλληλέγγυα κοινότητα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Η κυρία Στέβενς έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το μοναδικό αποτέλεσμα της μήνης συνόδου είναι 100.000 έξτρα θέσεις ε, στην οδό των Βαλκανίων. Αυτό είναι όλο. Η έξοδος αυτή μαζική προς τη Δυτική Ευρώπη και από οικονομικούς μετανάστες συνεχίζεται και με καλύτερο τρόπο και πιο οργανωμένα πλέον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να κάνει συμφωνίες για βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και κάνει και τέτοιες ε, προτάσεις για τις επαναπροωθήσεις, pushbacks, ε, αποθήσεις που επιτρέπονται με βάση τη ε, διεθνή πρακτική και το διεθνές δίκαιο. Αλλά δεν έχουμε ποτέ ε, κοιτάξει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Το 2015 ήρθαν 500.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και μόνο. Η ε, Τουρκία χρησιμοποιεί τώρα τους πρόσφυγες ε, για, ε, ως αντάλλαγμα για την κατάργηση θεώρησης διαβατηρίων ακόμα και για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να φυλάσσουμε καλύτερα τα ε, θαλάσσια σύνορα. Για ποιο λόγο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί ή δεν θέλει να φυλάσει τα εξωτερικά της σύνορα. Έχει το ηθικό χρέος ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει αυτή την πολιτική που προσελκύει τυχοδιώκτες στην Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζούμπερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κατά τις τελευταίες συναντήσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, δεν υπάρχει πλέον αλληλεγγύη. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του τελευταίου Συμβουλίου ε, αφορούν το πώς να εκδιώξουμε τους πρόσφυγες. Αυτό το είδαμε μέσα στα πλαίσια της καταστολής κατά των ανεπιθύμητων και λέμε ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό και με παράνομες κρατήσεις. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες όπως τους εγκληματίες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι έγινε στην ε, τσεχική δημοκρατία. Γνωρίζουμε επίσης τι γίνεται και με στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη χρήση στρατιωτικών μέσων για την απόθυση των προσφύγων. Θα πρέπει να μας πείτε τι συμβαίνει με αυτές τις στρατιωτικές ε, αποστολές επιτόπου. Η κυρία Ζολίγια, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής και του Συμβουλίου, στις 11 και 12 Νοεμβρίου θα μεταβείτε στη Βαλέτα για μία διάσκεψη κορυφής για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε όμως ότι μέσα στα πλαίσια της παράνομης ή νόμιμης μετανάστευσης θα γίνουν πολλές διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα κράτη-μέλη εμένουν στην στρατικοποίηση των συνόρων τους και σε συμφωνίες, αμφίβολες συμφωνίες με τους ε, γείτονες. Η εκμετάλλευση και η διακίνηση ε, στην ουσία ανετίθενται σε ε, διακινητές, αλλά δεν θα πρέπει να δώσουμε και στρατιωτική απάντηση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους μετανάστες και τους πρόσφυγες για να αποφύγουμε τα δράματα θα πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας και να ταχθούμε υπέρ της αλληλεγγύης. Μαχ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα τα συμπεράσματα και πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη. Είναι ο δίθεν ανθρωπισμός. Αυτοί που μιλήσατε και καταπολεμήσατε τις κυβερνήσεις της Συρίας και της Λιβύης ε, ενδιαφέρονταν ε, για τους ανθρώπους ή για να διώξετε πολιτικούς. Εσείς που ανοίξατε τις αγκάλες σας, τους μετανάστες και πρόσφυγες, θέλετε, το εννοείτε πραγματικά ή θέλετε να δείξετε πόσο καλοί είσαστε. Το Συμβούλιο λέει ότι θέλει να ενισχύσει τα εξωτερικά σύνορα, αλλά εσείς ψηφίσατε για την θύλαξη των ε, εξωτερικών σύνορων και αυτό είναι ένα ψευδοτρίκ το οποίο ε, είναι, μας δείχνει πόσο ε, δύσκολα αντιμετωπίζουν μια κατάσταση, δηλαδή ψευδούς ανθρωπισμού. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για την μετανάστευση από χώρες της Αφρικής. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση έμπρακτα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει δηλαδή να προβάλλουμε προστασία για αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται και να δημιουργήσουμε και ασφαλείς ζώνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο. Φαίνεται ότι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις ε, στην ουσία τρέχουν γύρω-γύρω χωρίς να κάνουν τίποτα. Ίσα-ίσα ε, επιδίδονται σε μια κατάσταση δημιουργίας χάους, όπου λέμε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Αυτό είπε και ο καγκελάριος Φάιμαν. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική ευθύνη και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους ανάλογα από το που προέρχονται. Αυτό προβάλλεται επί της ουσίας. Δυστυχώ Πόνς, ε, δυστυχώς δρούμε με μεγάλη καθυστέρηση εκεί όπου παίζονται ανθρώπινες ζωές. Στο Συμβούλιο μιλάμε για τα ίδια χωρίς να αλλάξει τίποτα. Το προσφυγικό γίνεται θεσμική κρίση. Τα κράτη-μέλη δεν ε, εφαρμόζουν τα μέτρα της Κομισιόν. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση ε, συμβιβασμού, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε τον πόλεμο. Δημιουργούμε νέα εσωτερικά τείχη και ελπίζουμε τρίτες χώρες να λύσουν το δικό μας πρόβλημα επιγόντως και ρίχνουμε την ευθύνη ημέν τους δε για αυτά που κάνουμε ή δεν κάνουμε. Το ερώτημα πολλών πολιτών είναι μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που βλέπουμε κάθε μέρα στις ειδήσει. Δυστυχώς δίνουμε το λόγο στους αντιευρωπαϊστές, δηλαδή το μίσος προς τους ξένους και τον εθνικισμό. Η προσφυγική κρίση ήταν ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα και τώρα γίνεται καθαρά πολιτικό. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν θέλουν να δεχτούν περισσότερους πρόσφυγες, αλλά δεν θέλουν να ασχοληθούν ούτε με τον πόλεμο. Δηλαδή, θέλετε όλοι οι άλλοι να ασχοληθούν και με τους πρόσφυγες και με τον πόλεμο. Εάν δεν κατανοήσουμε ότι ο πόλεμος που εξωθεί τους πρόσφυγες είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πόλεμος ε, κατά των Σύρων είναι και πρόβλημα και πόλεμος κατά της Ευρώπης, δεν θα επιλύσουμε το θέμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι πρόσφυγες ε, και εμείς οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουμε τον ίδιο πόλεμο, απλώς δεν το συνειδητοποιούμε. Βάιντεν Χόλτσερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία η Κομισιόν. Ήμουν επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα στο, στη Γευγελή, στο Πρέσεβο και στην Τάσα. Αν δείτε εκεί στους ανθρώπους, είναι εξαντλημένοι, είναι απεγνωσμένοι, είναι απελπισμένοι. Είναι μεγάλο το άγχος, ε, τεράστιο το στρες και ο ρυθμός. 7.000 και μόνο περνάνε στην Πάσα. Αυτό ε, είναι έξοδος λέγεται, δεν υπάρχει άλλη. Ε, λέξη για να το χαρακτηρίσει. Θα πρέπει να πέσουν οι ρυθμοί, να υπάρχει κάπως μια κατάσταση ήρεμη, να κατευναστεί. Χρειάζεται βοήθεια επίγουσα και γενναιόδορη, έτσι ώστε τα hot spots, τα κέντρα καταγραφής ε, στα εξωτερικά σύνορα να είναι αποτελεσματικά και να κάνουν τη δουλειά τους. Και να έχουμε ε, υποδομές στα Βαλκάνια, σε αυτή την οδό που να αντέξουν το χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κρίπεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μία από τις προτεραιότητες σε αυτή την κρίση είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων. Μία πραγματική συνεργασία θα μπορούσε να αφορά ε, συγκεκριμένες δυνάμεις ενίσχυσης στην Ουγγαρία Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και η βοήθεια προς την Τουρκία έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία μιλάει για επιτάχυνση της διαδικασίας προσχώρησης, αλλά παράλληλα δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα ε, ενός κράτους που θέλει να προσχωρήσει. Η καγκελάριος Μέρκελ μίλησε για ένα πλαίσιο συνεργασίας και για άνοιγμα νέων κεφαλαίων. Δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξουμε τις προσφυγικές ροές, αλλά δεν αλλάζουμε καθόλου τη στάση μας. Πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε. Κυρία Σακόρα, ένα λεπτό. Κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέμαι για πόσα χρόνια ακόμα θα συζητάνε Επιτροπή και Συμβούλιο για το πώ θα αντιμετωπίσουν αυτή τη χωρί προηγούμενο ανθρωπιστική κρίση. Απέναντι σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, την τραγική πραγματικότητα, παρακολουθήσαμε τη χθεσινή φάρσα τη σημερινή Συνόδου Κορυφή. Τα συμπεράσματα που συζητάμε σήμερα δεν αντέχουν σε καμιά κριτική και αποτελούν ύβρι για τα εκατομμύρια των προσφύγων, για του χιλιάδε νεκρού, αλλά φυσικά και για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και η ανθρωπιστική κρίση αποκάλυψε τη γνία τη ευρωπαϊκή πολιτική η γερμανία απροκάλυπτα θέλει να μετατρέψει τον νότο και ειδικά την ελλάδα σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης ενισχύοντας έτσι πολιτικές κλειστών συνόρων μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση. παράλληλα παίζει επικίνδυνα παιχνίδια αποσταθεροποίησης με την τουρκία σε βάρος τόσο της ευρωπαϊκής πολιτικής διερεύνησης όσο και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. μόνο όποιος εθελοτυφλεί δεν αντιλαμβάνεται ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αποκαλύπτεται τα σταθρά θεμέλια του το έχω ξαναπεί λοιπόν ότι η ανθρωπιστική κρίση ξεπερνάει κατά πολύ το δίλημα του ποια ευρώπη θέλουμε. αν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική απλά δεν θα υπάρχει ευρώπη. Ευχαριστούμε. Κύριε Άτκινσον για ένα λεπτό. Η αριστερά και ο κύριος Πιτέλα σήμερα έφτασαν σε ένα καινούργιο ναδύρ. Ο κύριος Σούλτς απ' την άλλη λέει ότι δεν πρέπει να προασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα. Πρέπει ο λαός της Βρετανίας να φύγει από εδώ μέσα εγκαίρος. Ο κύριε Γιούνκερ, όποτε έχετε μια αμφιβολία να οργανώνετε μια διάσκεψη κορυφής. Έρχεται εκπρόσωπος της Προεδρίας να μας μιλήσει για τους ε, πρόσφυγες, αλλά κανείς δεν έρχεται στο Λουξεμβούργο ως πρόσφυξ οι ροές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διπλασιαστεί και εγώ λέω ότι δεν είναι πρόσφυγες αλλά οικονομικοί μετανάστες. Φαίνεται δεν υπήρξε μετάφραση στα γαλλικά. Δεν πειράζει, εγώ θα συνεχίσω γιατί μιλάω για τους Βρετανούς. Λοιπόν, δεν είναι πρόσφυγες αλλά οικονομικοί μετανάστες και το κύριο τους μέλημα δεν είναι η ασφάλεια αλλά οικονομικό κέρδος. Χθε ήμουν στο Eurostar και ε, ήταν εκεί μέσα ε, πάνω στις ράγες ορισμένοι μετανάστες δεν τους συνέλαβαν οι αρχές δεν έκαναν τίποτα και αυτό είναι λάθος γι' αυτό θα καταστραφεί αργά ή γρήγορα αυτό το μέρος η Ευρώπη δηλαδή ο κύριος Μπρόκ ε, έχει μπλε κάρτα ε, όχι έχουμε ψηφοφορίες δεν θέλω να σας καθυστερήσω δεν περίμενα και τίποτα άλλο όπως σας λέει ο πρόεδρος Κύριε Μπροκ, ο διάλογος ήταν μεταξύ ε, της εξαιρέτης συναδέλφου και του Βρετανικού ε, Ακροατηρίου και ψηφοφόρων. Ας μην αναμειγνιόμαστε εμείς σε τέτοια πράγματα. Η κυρία Γκαρντίνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σαν Ιταλίδα θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ξεχάσατε την Ιταλία. Δεν την αναφέρατε και εμείς έχουμε να κάνουμε με μικρές αψιμαχίες ε, μπροστά στο ευμέγεθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. αντιμετωπίζουμε. Όπως είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, τα μέσα που διαθέτουμε δεν είναι απεριόριστα. Ε, άρα ε, τι μπορούμε να πούμε, ούτε η αλληλεγγύη μας δεν πρέπει να είναι απεριόριστη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα κατεπηγόντως με βάση αυτά που συμφωνήθηκαν. Ακόμα κι αν κερδίσει αυτός που λέει στεγανά σύνορα ή εκείνος που λέει αλληλεγγύη, η Ευρώπη θα κατακαιρματιστεί, γιατί αυτό είναι ένα από τα βήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή το κατεπήγον ζήτημα. Αν δούμε όμως το γεωπολιτικό σύστημα, από πού φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουμε πώς πρέπει να εργαστούμε, έτσι ώστε οι μετανάστες να μπορούν να ζήσουν εκεί από όπου προέρχονται, να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να απεριμόνονται περιοχές που απεριμόνονται όχι λόγω κλιματικών αλλαγών, αλλά για πολιτιστικούς λόγους. Ένας μεγάλος Ιταλός, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη, το 60 ήταν προφήτης και μίλησε για τον Αλή με τα ε, μπλε μάτια θα είναι πολλοί άνθρωποι που θα έρθουν στο Κροτόνε, στο Πάλμι, θα είναι ρακένδυτοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν στις ακτές μας. Ήταν μεγάλος προφήτης αυτός ο άνθρωπος στη δεκαετία του 60. Ας δώσουμε σίγουρες και μόνιμες απαντήσεις. Νίτερ Μίλλερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε τα 17 σημεία για τα Δυτικά Βαλκάνια, αυτός ο δικός χάρτης είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Σημαίνει ότι μια κοινή Ευρώπη που βασίζεται στην αλληλεγγύη μπορεί να ε, επιζήσει με κοινά σύνορα. Δεν θα πρέπει να προβάλλουμε φράκτες αποκλειστικά και τον εγωισμό μας. Φτάσαμε σε αποτελέσματα την προηγούμενη Κυριακή και δεν μιλώ μόνο για επιχειρήσεις στα σύνορα. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την ενσωμάτωση τάχιστα των προσφύγων. Χρειάζεται ολοκλήρωση, ενσωμάτωση και όχι ψευδοενσωμάτωση. Πρέπει να μάθουν τη γλώσσα μας αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό χρειαζόμαστε πολλά χρήματα. Ας μην δημιουργούμε ένα κλίμα φόβου. Ας υπάρξει μία πολιτική ένταξης και αυτό ας το κάνουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει κοινή πολιτική, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκάλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η μεταναστευτική κρίση είναι μόνιμο θέμα στην ατζέντα μας. Παράλληλα υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη πίεση προς την Ευρώπη και εμείς παραμένουμε αναποφάσιστοι. Χρειαζόμαστε καινοτόμο δράση και ευθύνη έτσι ώστε η αλληλεγγύη να μεταφραστεί σε πράξεις. Γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε την πολιτική των ανοιχτών συνόρων θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η διάσκεψη κορυφής έδειξε ότι αντιμετωπίσαμε τα πλέον βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Δεν μπορούμε να ομφαλοσκοπούμε. Ο δρόμος των Βαλκανίων είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κατάσταση ολοένα και θα επιδεινώνεται. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν από τον Αύγουστο. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας στην ουσία λιδωρήθηκε για τη στάση του σε σχέση με την ανύψωση των τυχών και φυσικά θα πρέπει να γίνει καταγραφή των προσφύγων και των μεταναστών και δεν πρέπει να επιλέγουν πού θα ζητήσουν άσυλο. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα μέσα στην Ευρώπη, εκτός και αν υπερασπιστούμε τα εξωτερικά μας σύνορα και να πούμε στους ανθρώπους ναι μπορείτε να έρθετε, αλλά αυτή είναι η ποσόστοση. Έτσι θα υπερασπιστούμε το, και το σύστημα Σέγγεν. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους σε αυτούς τους καταβλισμούς. Πολλοί θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Και η διάσκεψη της Μαδρίτης του ΕΛΚ το τόνισε. Μιλώντα γι' αυτό το θέμα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το δρόμο χρησιμοποίησαν και, χρησιμοποίησε και ο στρατός, οι μεγάλες στρατιές που πήγαν να κατακτήσουν τη Βιέννη. Η κυρία Γκαρθία. Μιλάμε για άμεση αντίδραση. Δεν ξέρω τι σημαίνει για σας αυτό. Μας οχλεί πλέον η υποκρισία. Μιλάμε για αλληλεγγύη. Το λένε πολλά μέλη, ενώ οι κυβερνήσεις τους δρούν ολέθρια. Γιατί εδώ και ένα μήνα μιλήσαμε για κλίδα κατανομής των προσφύγων και χτες η κυβέρνηση του κυρίου Ραχώη είπε ότι θα στείλει ορισμένους υπαλλήλους για να υποδεχτούν τους 50 πρώτους ε, πρόσφυγες. Αν δεν μιλούσαμε για κάτι τόσο σημαντικό θα έλεγα πρόκειται για αστείο. Η εικόνα του κυρίου Όρμπαν στο ΕΛΚ στη Μαδρίτη, ο οποίος ε, στην ουσία καταχειροκροτήθηκε μέσα στα πλαίσια των αντιδραστικών του δηλώσεων, αφήνει ένα μήνυμα ότι παίζουμε με τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων. Η κυρία Σουίτσα για ένα μισή λεπτό. mene kao hrvaticu brine situacija kako... Ως κροάτισα ανησυχώ για την κατάσταση και για το πώς μπορούν να συνδυαστούν όλοι οι εθνικοί εγωισμοί με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Είναι καλό που την Κυριακή όλοι οι αρχηγοί των Βαλκανικών χωρών συναντήθηκαν. Δυστυχώς έχει φύγει εδώ ο κύριος Γιονκέρα, αλλά αυτοί οι αρχηγοί κρατών δεν μπόρεσαν να οργανώσουν μόνοι τους μια τέτοια συνάντηση διότι κάθε χώρα μόνη της προφανώς δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει το πρόβλημα και είναι καλό να το οργανώσουν οι οργανισμοί, οι θεσμοί. Συμφωνώ με τον κύριο Γκονζάλες ότι ο πόλεμος κατά της Συρίας είναι πόλεμος κατά της Ένωσης. Επίσης πρέπει να στηρίξουμε την Τουρκία γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Έρχεται ο χειμώνα και αν δεν αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις που πήραμε δεν θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να κάνουν τίποτα. Πρέπει να εφαρμόσουν τις αποφάσεις αλλιώς θα καταλήξουμε στο χάος και ως πολιτικοί έχουμε καθήκον και αυτό περιμένουν οι πολίτες να λύσουμε τα προβλήματα πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε, να καταλάβουμε την δυνατότητα πραγματικής αποσταθεροποίησης του ευρωπαϊκού οράματος. Μωράης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρέπει πράγματι να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και είναι σοβαρό ό,τι πολιτικές απόψεις και να έχουμε να μην παρατήσουμε το ευρωπαϊκό όραμα. Γι' αυτό το λόγο ο Επίτροπος Αβραμόπουλος και η Επιτροπή Προπολογισμών θα μας συναντήσουν λίγο με, συνομιλήσουν μαζί μας δύο λίγα λεπτά μετά την ψηφοφορία. Νόθηκε η διάσκεψη των Δυτικών Βαλκανίων παρά τις επικρίσεις που ακούστηκαν. Πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα του χάους και επειδή έρχεται ο χειμώνας θα αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερους θανάτους. Πρέπει να κάνουμε κάτι και αυτό σημαίνει ότι το κοινοβούλιο μα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Μετά τις συζητήσει να αρχίσει η πραγματική δουλειά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να ε, λειτουργήσουν τα hot spots και τα κέντρα υποδοχής. Αν αυτά λειτουργήσουν σωστά, τότε αφού έγινε αυτό επιτεύχθηκε και στο παρελθόν μπορεί να επιτευχθεί και στο μέλλον. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ο κύριος Κεφαλογιάννης παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Το Συμβούλιο υπήρξε μια σημαντική συνάντηση. Υπήρξε αύξηση της δυνατότητας υποδοχής προσφύγων σε 100.000 σε όλο το μήκος του Βαλκανικού διαδρόμου από τα ελληνικά σύνορα ως τα σύνορα της Αυστρίας με τη Γερμανία. Μόνο στην Ελλάδα δόθηκε η δυνατότητα, δέχτηκε δηλαδή η Ελλάδα, να έχει παραπάνω 50.000 πρόσφυγες και να δημιουργήσει κομβικά σημεία hot spots για το κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης των προσφύγων. Υποδοχή λοιπόν 30.000 προσφύγων και πρόβλεψη για άλλους 20.000 πρόσφυγες με επιδότηση ενοικίου και την υποστήριξη της ύπατης αρμοστίας του οργανισμού ηνωμένων εθνών. αυτό που έλειπε από τη συνάντηση είναι η τουρκία. είναι η κοινή δράση το κοινό πρόγραμμα δράσης με την τουρκία μακριά από ανατολίτικα παζάρια και κυρίως εν ώψη εκλογών στην τουρκία. έλειπε η συνάντηση με τα αφρικανικά κράτη. είναι σημαντικό που ο κύριος Τούς και ο κύριος γιούνκερ ανακοίνωσαν τη συνάντηση στη βαλέτα νομίζω ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην κοινή μας προσπάθεια και κυρίως λείπουν τα πλούσια αραβικά κράτη με εξαίρεση το λίβανο και την ιορδανία. μόνο στην σαουδική αραβία κυρίες και κύριοι συνάδελφοι υπάρχουν, εγκαταστάσει εγκαταστάσεις με τέντες έτοιμες για τρία εκατομμύρια πρόσφυγες. κρινόμαστε όλοι κρίνεται η ευρωπαϊκή ένωση κρινόμαστε εάν πράξαμε το χρέο μα απέναντι στι προσπίσει. Κύριε Περβάς ε, Μπερέζ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια κρίση και έχουμε την εντύπωση ότι την υφίσταται, δεν την ελέγχει. Ποιος ενδιαφέρεται για την κατάσταση στη Συρία, ποιος λέει ότι με μαζικές αυτές μεταναστευτικές ροές συμβαίνουν επειδή προοδεύει τον τάες στη Συρία. Ποιος λέει ότι δεν θα υπάρξει λύση με τον κύριο Ασάντ. Ποιος λέει ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τις σχέσεις Ένωσης Ρωσίας. Κύριε Πρόεδρε, πέστε στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι πρέπει κάτι να κάνει, αλλιώς μεταξύ μας δεν θα υπάρχουν πραγματικές σχέσεις αλληλεγγύης παρά μόνο αλληλεξάρτησης όπως έγινε με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση στραβά, όπως έγινε με το Σέγγεν χωρίς πολιτική ασύλου, χωρίς ευρωπαϊκή υπηρεσία για τους πρόσφυγες, χωρίς εξωτερική προστασία των συνόρων. Ζητώ από τον πρόεδρο της Κομισιόν να τα συνδυάσει όλα αυτά και να κάνει, αναλάβει μία πρωτοβουλία που να λύνει πράγματι αυτά τα προβλήματα ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να επιστρέψει. λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή ε, τι μας κάνει, μας βάζει μπροστά μας ένα καθρέφτη. Αν δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να δούνε τον άνθρωπο μέσα σε αυτή τη μάζα ανθρώπων, τότε τι να πούμε. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να είμαστε ε, ψυχροί προς τους ανθρώπους, ανάλγητοι, που είναι ε, πρόσφυγες και χρειάζεται αλληλεγγύη με τις χώρες που υποδέχονται τους περισσότερους. Και αυτή η σαφήνεια είναι να πεις με κάθε ειλικρίνεια ότι κοίτα εσύ δεν χρειάζεσαι την προστασία μας και με τρόπο αξιοπρεπή και κανονικό να οργανώσουμε την αποχώρησή του. Αυτό θα κοστίσει και κόπο και ε, χρόνο και χρήματα. Και όχι όπως κάνουν τα κράτη-μέλη που τάζουν διάφορα, δεσμεύονται και μετά δεν κάνουν τίποτα ε, και μετά προχωρούν και νομίζουν ότι είναι όλα δωρεάν. Ε, πού είναι η ανθρωπιά που ακούμε εδώ μεγάλα λόγια. Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να φυλάσσουμε τα σύνορά μας και γι' αυτό χαίρομαι που ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα φέρει γρήγορα πρόταση για ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Χαίρομαι και για τη συνεργασία που έχουμε και την οικονομική με τρίτε χώρε γειτονικέ. Βέβαια έχω τι αμφιβολίε μου κατά πόσο θα πρέπει να συνδεθεί αυτή η συζήτηση για του πρόσφυγε με τη συζήτηση για την ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α είμαστε ειλικρινεί και σαφεί μεταξύ μα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Νταλή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η διάσκεψη κορυφής έδειξε τις εντάσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια στιγμή που υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και μιλάει με μια φωνή. Η διάσκεψη της Βαλέτας είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει επικοδομητική συνάντηση με την Αφρικανική Ένωση για να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Οι μεταναστευτικές ροές υπάρχουν εξαιτίας της φτώχειας, της εμπόλυμες κατάστασης και της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει να παρασχεθεί βοήθεια και να δοθεί και να γίνουν πραγματικές αλλαγές. Θα πρέπει οι πολίτες να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλήσει με μία ενιαία φωνή, αν θέλουμε να προβούμε σε αλλαγές. Ρανζέλ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και τη συνάντηση που έγινε το Σαββατοκύριακο με τις χώρες, τις 11 χώρες που έχουν σχέση με τα Βαλκάνια και που δέχονται πρόσφυγες θα πρέπει να μας οδηγήσει στο ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή ευθύνη και όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Όλοι θα πρέπει να υποδεχτούμε πρόσφυγες, είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό και θα πρέπει να παρασχεθεί και οικονομική βοήθεια και σε εκείνους που βρίσκονται εκτός συνόρων, των δικών μας δηλαδή συνόρων. Θα πρέπει να υπάρχει μία αλληλεγγύη με συγκεκριμένα κριτήρια. Θα πρέπει να μην συγχαίουμε τους πρόσφυγες με τους μετανάστες. Θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση ιδιαίτερα στα hot spots, στα σημεία υποδοχής και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που βρίσκονται στην ε, εμπροστοφυλακή, είτε είναι κράτη-μέλη είτε όχι. Πρόκειται για κοινή μας ευθύνη και θα πρέπει να την αναθέσουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Από τη δική μας άποψη έχει μεγάλη σημασία να προβούμε και σε μια εργασία πρόληψης, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική ιδιαίτερα στα έφλεκτα σημεία όπου χρειάζεται μία κατεπίγουσα απάντηση και μιλώ για την υποσαχάρια Αφρική. Η κυρία Μίτσι, για ένα λεπτό. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η μετανάστευση είναι σύμπτωμα και όχι το αίτιο του προβλήματος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα αίτια και να τα αντιμετωπίσουμε, δηλαδή την εμπόλεμη κατάσταση, τις ε, τρομοκρατικές ενέργειες και τη βία. Αυτά είναι μερικά από τα ενάυσματα και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και να φτάσουμε σε μια διεθνή λύση στην κρίση της ε, μετανάστευσης, που μπορεί να δοθεί αν αντιμετωπίσουμε τα θεμελιώδη αίτια της ε, κρίσης. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αφορμή στη χώρα μου στη Μάλτα, στη Βαλέτα, τη διάσκεψη δηλαδή με την Αφρικανική Ένωση για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις για να μην φεύγουν από την πατρίδα τους ε, οι άνθρωποι αυτοί δεν υπάρχει ενιαία λύση, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ένα μέλλον σε αυτούς τους ανθρώπους και να μην διακινδυνεύουν τη ζωή τους ε, αποζητώντας μία αξιοπρεπή ζωή. Χρειαζόμαστε μακροχρόνια στρατηγική. Wilmot. Εξ του Εργατικού Κόμματος ε, δέχομαι τη συνεργασία με την Τουρκία για να διαχειριστούμε καλύτερα την Τουρκία. Ακούσαμε τους κοινικούς που μιλάνε ότι δεν θα φτάσουν, για το γεγονός ότι δεν θα φτάσουν σε λύσεις, αλλά θα χρησιμοποιήσουν στρατηγικά αυτό το πολιτικό παιχνίδι. Τώρα μιλάμε για απόδοση, για λύση. Πρόκειται για ένα μεγάλο εφιάλτη όλων αυτών των οικογενειών που διανύουν μίλη με μίλη αυτή την τεράστια απόσταση για να έχουν αξιοπρεπή ζωή. Δεν είναι πολιτικό παιχνίδι, πρόκειται για αξιοπρέπεια Μιλάμε και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για το δημοψήφισμα. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον Πρωθυπουργό Κάμερον ότι δεν υπάρχει πια καθυστέρηση, δεν μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση. Η Βρετανία θα πρέπει να έχει το μέλλον που της αξίζει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήρε για ένα λεπτό. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, ε, δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δέσμευσή της να βρεθούν πρακτικές λύσεις σε αυτή τη τεράστια πρόκληση που όλοι αντιμετωπίζουμε. Καλωσορίζω το πρόγραμμα δράση που από κοινού εκπονήθηκε με την Τουρκία, καθώ η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται μία την άλλη για να μοιραστούν το βάρο και να δώσουν ασφαλέ καταφύγιο για τόσου πολλού ανθρώπου που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την οικονομική βοήθεια, ε, επανεκατάσταση, ε, ε, αποτελεσματική επιστροφή των μεταναστών και καταπολέμηση των διακινητών αρνούμε να δεχτώ τη σύνδεση με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν καμία σχέση τα θέματα. Ε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την έκθεση πρόοδου. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να σταματήσει να εκφράζει την κριτική της ε, για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώπιον σημαντικών εκλογών. Δεν θα πρέπει να στέλνουμε λάθο μηνύματα. Να συνεχίσουμε να εκφράζουμε την ανησυχία μα για την ελευθεροτυπία και την κατάσταση τη κουρδική μειονότητα. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Τόγια, για ένα λεπτό. Εγώ ξεκινώ από τα λόγια του Προέδρου Γιούνκερ που είπε ότι τα, πρόβλημα, τα προβλήματα των μεν είναι τα προβλήματα και των δε. Αυτό ισχύει για κάθε κοινωνία και για τα θεσμικά όργανα. Η Ευρώπη θα σταθεί στα πόδια της αν βασιστεί στην αλληλεγγύη, γιατί σήμερα μιλάμε για αυτούς τους πρόσφυγες, αύριο θα είναι άλλοι. Αν δεν υπάρχει ενωτική προσέγγιση, δεν θα πρέπει να κάνουμε λάθη όπως κάναμε έναντι της Σλοβενίας, έναντι της Ελλάδας κλπ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που ζουν μέσα στη λάσπη, μέσα στα έλλη, αυτοί που αντιμετώπισαν τον το ήλιο της Μεσογείου το καλοκαίρι. Κύριε Τούσκ, θα πρέπει να μας καθοδηγήσετε έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται με τις δράσεις μας για να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις θα πρέπει, ε, όπως είπε και ο κύριος Πιτέλα, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Αφρικανική Ένωση. Να, συνεργαστεί και, ο, και να συνεργαστούν και οι χώρες του Περσικού κόλπου για να αντιμετωπίσουμε την ε, αποσταθεροποίηση που υπάρχει. Πιτσούλα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη Κροατία είχαμε 250.000 μετανάστες που έφτασαν στην Κροατία. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση χωρίς ε, στρατικοποίηση των ε, συνόρων. Δεν τους ε, οθήσαμε να πρέπει να διασχίσουν ποτάμια υπό εκτρές συνθήκες όπως, όπως προαναφέρθηκε. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι έχουμε 10.000 ε, λέψεις καθημερινά και δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τα Βαλκάνια. Θα πρέπει να λύσουμε και το θέμα των εξωτερικών μας σύνορων. Ας στραφούμε στη συνεργασία και όχι στο να λιδωρούμε ο ένας τον άλλον. Διαφορετικά, οι χώρες που εκτίθενται θα δεν μπορούν παρά να αντιμετωπίσουν θέμα ασφάλειας. Ο κύριος Κύρκος έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προχθέ μα παρουσιάστηκε η Συμφωνία των 19 Σημείων που είναι πάρα πολύ σημαντική αν τελικά καταφέρει να υλοποιηθεί γιατί οι δειλές και αργοπορημένες απαντήσεις είναι αυτές που εξέθρεψαν το πρόβλημα στις κοινωνίες υποδοχής που κάνουν την ξενοφοβία να φουντώνει. Όμως πρέπει πάλι να σας προειδοποιήσουμε. Χωρίς μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, οι πρόσφυγες δεν θα κάτσουν ούτε τρεις μέρες στα κέντρα υποδοχής, αν αυτά μπορεί να γίνουν φυλακές. Και χωρίς ε, αιτήσει ασύλου σε ευρωπαϊκά γραφεία στην Τουρκία και μόνιμους δρόμους, ασφαλείς δρόμους προσέγγισης, δεν θα σταματήσουν οι πνιγμοί στο Αιγαίο. Και υπάρχει μία απάντηση. Η Τήλος, ένα μικρό νησί χαμένο στον Ανατολικό Αιγαίο, ξεχασμένο από Θεό και κυβέρνηση, χωρίς γιατρό και δάσκαλο. Όμως η Τήλος ζήτησε 100 οικογένειες Σύρων προσφύγων να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί. Γιατί εκεί υπάρχει ηγεσία, εκεί υπάρχει μία κοινοτάρξη η οποία δείχνει το δρόμο της αλληλεγγύης και οι κάτοικοι οργανώνονται και ακολουθούν. Ευχαριστώ. Ακολουθεί τώρα η διαδικασία Κατσιάη. Επτά συναδέλφους θα αφήσω να μιλήσουν. Έχουμε άπειρες αιτήσει που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τις λάβουμε υπόψη. Η κυρία Βόζεμπερκ, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Στη Μικρή Σύνοδο Κορυφή την 25 Δεκάτου αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η φιλοξενία μέχρι τέλο του έτου στην Ελλάδα 30.000 προσφύγων και άλλων 20.000 με επιδότηση ενοικίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια χώρα που βρίσκεται έκτη χρονιά σε οικονομική κρίση με εφιαλτική ανεργία, ούτε τροφή, ούτε ένδυση, ούτε περίθαλψη είναι δυνατό να παρασχεθεί στου ανθρώπου αυτού, αλλά μόνο προβλήματα με απρόβλεπτε συνέπειε. Η απόφαση αυτή άλλωστε ακυρώνει στην αλλάξει το μέτρο της μετεγκατάστασης 64.400 προσφύγων από την ελλάδα που ισχύει από τον περασμένο οκτώβριο. σοβαρή προσέγγιση του προσφυγικού σημαίνει υπεύθυνη συνεργασία με την τουρκία που είναι χώρα διέλευσης ώστε να τηρηθούν οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν υπογραφεί αλλά κυρίως να ελεγχθούν αποτελεσματικά τα δίκτυα των λανθρεμπόρων που εκμεταλλεύονται τα κύματα των μεταναστών προς την ευρώπη. διαφορετικά το προσφυγικό θέμα κινδυνεύει να αποδειχθεί μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία καταρχάς, σταματήστε τις ανοησίες για το πραξικόπημα στην ε, Πορτογαλία. Σημείωσε αυτό που είπε ο κύριος Βέμπερ ότι ανησύχησε για την κατάσταση. Αλλά ε, στη χώρα μου είναι τελείως νόμιμο αυτό μετά τις εκλογές. Από ό,τι φαίνεται δεν ανησυχεί για μια ξενόφοβη αντιευρωπαϊκή ακροδεξιά κυβέρνηση στην Πολωνία που έτσι διαγράφεται. Τουλάχιστον στην Πορτογαλία εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχόμαστε πρόσφυγες. Ε, όλες ε, οι αρχές ε, που ενέχονται στην υποδοχή. Αλλά το θέμα είναι ότι η διαδικασία επανεκατάστασης δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έρχονται οι άνθρωποι. Τουλάχιστον στη Σύνοδο της Βαλέτας ελπίζω να είναι η ευκαιρία για όλους τους ηγέτες να καταλάβουν τι έχουν ακούσε εδώ και τι είπα, ότι αν δεν αφήσουμε νόμιμες και ασφαλείς οδού για πρόσφυγες και μετανάστες θα εξακολουθούν να πέφτουν στα νύχια και να τροφοδοτούν αυτές τις εγκληματικέ συμμορίες. Και ούτε πρόκειται να τελειώσει η σύραξη στη Συρία, στη Λιβύη, ούτε να ιτηθούν οι τρομοκράτες στο Ιράκ και τη Συρία. Ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κακό στη ρίζα του. Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι. Δεν είναι προσφυγική κρίση, είναι πραγματικά ευρωπαϊκή κρίση, διότι αποτυγχάνουμε να προστατεύσουμε τους απροστάτευτους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι για τη συμφωνία της Κυριακής γιατί θα επιτρέψει στους πρόσφυγες να υποφέρουν λιγότερο και θα βοηθήσει τις χώρες υποδοχής και μετάβασης να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα όπως η χώρα μου η Κροατία που, από την οποία πέρασαν πάνω από 300.000 τελευταία. Δεν μπορεί όμως να απαγορευτεί η πρόσβαση στην Ένωση των Προσφύγων εκτός δια της βίας. Ελπίζω να βρεθεί μια ειρηνική λύση και μια μακροπρόθεσμη λύση για να βρεθεί μια λύση της κρίσης και στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Δυστυχώς όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το σκέφτεται καν αυτό. Κύριος Χατζηγεωργίου παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακολούθησα όλη τη συζήτηση των τριών περίπου ωρών. Με όλη την ειλικρίνεια σας λέω ότι αν ήμουν πρόσφυγας, ένας μετανάστης και άκουγα αυτή τη συζήτηση, κυριολεκτικά θα προσπαθούσα να βρω το δρόμο προς το Αιγαίο να πάω να αυτοκτονήσω. Από τις ανέξοδες ρητορικές υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων μέχρι την ομιλία του κυρίου Juncker, ο οποίος δεν παρέθεσε καμία ουσιαστική πρόταση άμεσης επίλυσης του προβλήματος. Θα πω και δύο λέξεις για την Τουρκία. Κατανοώ πλήρως την διάθεση συνεργασίας. Αλλά από τη διάθεση συνεργασίας μέχρι το να πάμε να λέμε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα μετά από την βομβιστική επίθεση, για να μην αναφέρω τους εκατοντάδες άλλους νεκρούς άλλων βομβιστικών ενεργειών ή επιθέσεων της Τουρκίας ενάντια στους Κούρδους, την, την εκατόμβη των εκατόν νεκρών στην άγκυρα να ονομάζουμε αυτή τη χώρα ασφαλή προκειμένου να διώξουμε το πρόβλημα από τη δική μας αυλή πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι παρεμβάσεις των Πρόεδρων Τούσκ και Γιούνκερ μας εξηγούν την αλήθεια που είναι η υπαρξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τους πολιτικούς. Μας σκανδαλίζουν οι διαμάχες στα σύνορα μεταξύ κρατών ε, μελών. Ακούμε και πώς διαπληκτίζονται εδώ μέσα οι πολιτικές ομάδες. Αλλά το πραγματικό σκάνδαλο δεν είναι στα Βαλκάνια, αλλά στη Δυτική Ευρώπη, στα μεγάλα και ισχυρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός που αποτυγχάνει δεν είναι Ευρώπη των 28, αλλά Ευρώπη των 15. συμφωνούμε για τα κέντρα καταγραφής, αλλά είναι μόνο αυτό, είναι μόνο 5% του προβλήματος. Δεν ακούσαμε ακόμα το μήνυμα που μας στέλνουν οι, οι πρόσφυγες. It's Europe, stupid. Η Ευρώπη είναι το θέμα. θα εκρίνουμε τώρα ακτοφυλακή, σύνοροφυλακή, ε, καταβλισμούς σε Γαλλία, Γερμανία, ε, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο. Θα πρέπει υπεύθυνα να δράσουμε επιτέλους, Πρόεδρε. Η Ευρώπη είναι το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χωρίς μικρόφωνο. Ακούμε διάφορες κατηγορίες εδώ πέρα. Κέντρα καταγραφής, κέντρα υποδοχής, κοινή ε, ε όλα και να λόγια, κούφια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ικτρά απέτυχε. Έχει αποτύχει το Σέγγεν, τα εξωτερικά σύνορα. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Καταστροφή για την εθνική κυριαρχία. Πάνω από ένα εκατομμύριο παράνομα ρέουν οι πρόσφυγες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξέλεγκτα και χωρίς καταγραφή. Πρόκειται για επέλαση, για κατοχή. 70 με 80% είναι νέοι άνδρες ε, που ψάχνουν την τύχη τους στη Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία κτλ. Δεν είναι απορία άξιο. Στη Συρία ξέρετε πόσο παίρνει ένας πανεπιστημιακός ή στο Αφγανιστάν. είναι χιονοστιβάδα αυτό που μας έρχεται και τα λόγια δεν βοηθούν. Χρειάζονται έργα, σταράτα και ξεκάθαρα. Ο κύριος Κούκα. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από την αρχή της κρίσης της μετανάστευσης έκανα έκκληση στους αρχηγούς Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, συμπεριλάβουν τα Δυτικά Βαλκάνια στη λύση του ζητήματος, γιατί χρησιμοποιούν αυτό τον ε, βαλκανικό διάβλο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα τρόπο πιο στενής συνεργασίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για να ε, αποσύσουμε και οποιαδήποτε μεταγενέστερη κρίση. Δυστυχώς η απάντησή μας ήρθε πολύ αργά. Χαίρομαι, η σκέψη της αντιμετώπισε το ζήτημα αυτό για άμεση δράση έναντι του πολέμου. Για να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές θα πρέπει να καταπολύσουμε και τους διακινητές ανθρώπων και να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια και κοινή διαχείριση πληροφοριών. Έτσι μπορούμε να προετοιμάσουμε αυτές τις χώρες καλύτερα για μελλοντική συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι πολύ ευχάριστο να μιλώ αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ όμως που μου δίνετε το λόγο. Εκτιμώ τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ως προς την εξέβρεση μιας λύσης στο προσφυγικό θα πρέπει να επικρίνουμε και τη στάση ορισμένων κρατών μελών που δεν ήταν έτοιμα να επιλύσουν ή να αντιμετωπίσουν την ε, κρίση. Θα ήθελα να πω προς τον ε, Επίτροπο ότι αυτό που έχει σημασία είναι η, και η ριζοσπαστικοποίηση και στα κράτη-μέλη που μόλις ε, βλέπουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές διαδηλώσεις αυτών των ακραίων δυνάμεων που δυστυχώς επιτίθενται και κατά των καταβλισμών. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τα κράτη-μέλη τα ίδια να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες για να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτό τον εθνικισμό στις χώρες. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρακαλούσα να καθέστε στις θέσεις σας. Meine Κυρίες και κύριοι, οι υπόλοιποι συνάδελφοι ε, που έχουν ακόμα ιδιωτικέ συνομιλίες και τις συνεχίζουν στην Ολομέλεια, καλό θα ήταν να καθίσουν στις θέσεις Θα ήταν πολύ ευγενικό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι δέκα τελευταίοι ομιλητές ε, ακούστηκαν από τον παραμικρό Ποια είναι η κοινοβουλευτική συζήτηση. Θα πρέπει οι συνάδελφοι να μπορούν να μιλούν και οι υπόλοιποι να τους ακούνε. Στους τελευταίους δέκα ομιλητές σίγουρα δεν συνέβη κάτι τέτοιο, μπορώ να σας το πω. Και το θεωρώ άδικο. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Επίτροπο. Παρακαλώ κύριε Βραμόπουλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι του Κοινοβουλίου, σήμερα ο πρόεδρος Γιούνκερ έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα για τη δραστηριότητα και στήριξη της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων. Αναλάβαμε δέσμευση και σημείωσα ότι υπήρξε και πολύ στεναρή στήριξη από εσά. Σχεδόν ομόφωνα. Χρειαζόμαστε τέτοια στήριξη από το Κοινοβούλιο και αυτά που πετύχαμε μέχρι τώρα οφείλονται σε αυτή τη στήριξη. Επίσης, χρειαζόμαστε από διάφορα κράτη μέσα και έξω της Ένωσης τέτοια στήριξη. Η μήνυ διάσκεψη της Κυριακής ήταν θετική, διότι οι χώρες που βρίσκονται πάνω στο δρόμο των μεταναστευτικών ή προσφυγικών ροών προσήλθαν και συζήτησαν και άρχισε ο διάλογος αλλά και όμως διάφορες χώρες χρησιμοποίησαν μόνο το εθνικό τους αφήγημα δεν υπάρχει ακόμα πλήρες ευρωπαϊκό πνεύμα συνεργασίας περισσότερη συνεργασία περισσότερη ελληνική περισσότερη ευθύνη χρειάζονται και φυσικά δράση, όχι μόνο δεσμεύσεις, όχι μόνο. Τώρα χρειάζεται η εφαρμογή, η πραγματική εφαρμογή. Αυτό είναι και το μήνυμα που πήρα από εσά σήμερα. Εφαρμογή και καλύτερη διαχείριση των συνόρων, προστασία σε όσους ζητούν άσυλο με πιο οργανωμένο τρόπο και συνεργασία με χώρες και εκτός Ένωσης. Ο ρόλος της Κομισιόν έχει αλλάξει με την κρίση αυτήν. Συνεχής επιτήρηση, εποπτεία και διάλογος χρειάζονται και πρωτοβουλίες με πιο στρατηγικό τρόπο. Γι' αυτό και το πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν θα πρέπει να δίνει ορισμένες απαντήσεις ο, για για όλα αυτά τα προβλήματα και τις μετακαταστάσεις των προσφύγων. Διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αποτύχει. Να μην ξεχνούμε ότι η κρίση των προσφύγων χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους στα εσωτερικά των διαφόρων κρατών μελών και στην κοινή γνώμη. Η μόνη λύση είναι να εξηγήσουμε στους πολίτες την ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση και αυτό σε διάφορα επίπεδα και να δείξουμε τον υποστηρικτικό ρόλο της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη και τις επηρεαζόμενες γειτονικέ χώρες. Εγώ είμαι πλήρως δεσμευμένος και έτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας και τις διάφορες χώρες έμεσα ή άμεσα με ευρωπαϊκές, αφρικανικές, ασιατικές χώρες και για την πολιτική των επιστροφών. Είχα σχεδιάσει να πάω αύριο στο Πακιστάν, αλλά λόγω του τρομερού σεισμού ανέβαλα το ταξίδι μου μία εβδομάδα. Θα πάω όμως, θα πάω. Και θα συζητήσω με τις πακιστανικές αρχές για την πολιτική των επιστροφών και των, τις δεσμεύσεις τους. Κύριοι βουλευτέ, η κρίση των προσφύγων είναι καταλήτης για περισσότερη Ευρώπη. Είναι μια δοκιμή για την Ευρώπη, δοκιμή αντοχής της αξιοπιστίας μας, των αρχών μας και των δυνατοτήτων που έχουν τα όργανα. Και αυτό κάνει η Κομισιόν, έχοντας βάλει την μετανάστευση στην κορυφή των προτεραιοτήτων της από την αρχή, αναλαμβάνοντας τις απαραίτητες όπως τη διάσκεψη της περασμένης Κυριακής ώστε να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο και αξία στις έννοιες της αλληλεγγύης και της ευθύνης και στηρίζοντας την ένωση, της, την ε, αξιοπιστία και της ίδιας της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κύριος Δόναλτ Τούσκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την κρίση αυτή. Η υλοποίησή τους δεν βαίνει με τους ταχύς ρυθμούς που χρειάζονται. Τώρα, οι κανονικές διαδικασίες σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αντικατασταθούν από έκτακτες επίγουσες καταστάσεις. Δυστυχώς αυτό δεν το έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει όλα τα κράτη-μέλη. Είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται να γίνει αυτό και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Λουξεμβουριανή Προεδρία είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ξεβρεθούν ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι εκείνοι που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής. Αλλά είμαστε και δίκαιοι. Οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα, στην ύπατη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες και σε άλλους οργανισμούς υπερβαίνουν τις μέχρι τώρα ε, δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Ξέρω ότι δεν είναι πιο εύκολη καιρή για τις κυβερνήσεις για να δαπανίσουν σήμερα ζεστό χρήμα, όπως μπορείτε να καταλαβαίνετε κι εσείς. Ίσως είναι η πιο δύσκολη απόφαση. Ας θυμηθούμε όμως για την επανεγκατάσταση ότι σήμερα είναι οκταπλάσιος ο αριθμός των θέσεων που προετοιμάζονται από τους πρόσφυγες εκείνους που θέλουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής. Πάντως θα πρέπει να έχουμε μια κοινή μέθοδο και ένα κοινό τρόπο και στόχο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Από την αρχή της παρούς κρίσης έχω υπογραμμίσει ότι σαφής μας στόχος θα πρέπει να είναι μια σημαντική συγκράτηση ε, του κύματος και των ροών αυτών της μετανάστευσης. Αλλά η άποψη που λέει ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο και η Ευρώπη θα πρέπει να δεχθεί όσους έρχονται εδώ, συνεχίζει να ακούγεται. Ακούστηκαν και σχόλια για τη συμπεριφορά προς τους πρόσφυγες ε, σε κάποια κράτη-μέλη από πλευράς των αστυνομικών αρχών. Ακούμε κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να τονίσω με κάθε στεναρό και κατηγορηματικό τρόπο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται όταν δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από χώρε που δεν υπάρχει ούτε διοίκηση ούτε αστυνομία καθόλου ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ένα προαπαιτούμενο. Την προστασία της δημόσιας τάξης και τη υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων. Και αυτό το γενικό σχόλιο αφορά όλα τα θέματα που σήμερα μας απασχολούν και συζητούμε στα πλαίσια της μεταναστευτικής ε, κρίσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τούσκ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση κυρίε και κύριοι. comes to the vote. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Πρώτο θέμα. Ο κύριος Ντάρθμον, θέλει το λόγο. Τι έχετε διαδικαστικό. I give the floor. Yes, I am. Ε, διαδικαστικό. Πρόεδρε. Είναι σωστό να συγχαίρουμε τον κύριο Ντόναλτ Τούσκ που αποφάσισε να παραιτηθεί ως Πρωθυπουργός της Πολωνίας πέρσι έτσι ώστε να αναλάβει την παρούσα θέση του ως πρόεδρος του Συμβουλίου και διακόπτε το ομιλητή. Αυτό δεν είναι διαδικαστικό, με συγχωρείτε. Γιατί. Um, we move on to Έκθεση Σικάρσκι. Σικέρσκι με ονομαστική κλίση, η οποία και αρχίζει. Πέρας. Πέρας.